παρομοίω Σήμερα αναφέρθηκε η συζήτηση ότι ενδεχομένω να ανακύψει παρεμφερέ πρόβλημα του χρόνου. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια κοινή συζήτηση για την δέσμη μέτρων για τους αερολιμένε. Αυτό το πακέτο ενέχει τρεις ε, διαφορετικές εκθέσεις. Η πρώτη είναι του Άρτουρ Ζασάντα για τις υπηρεσίες εδάφους ε, στους αερολιμένες της Ένωσης. Η δεύτερη ε, σχετίζεται με την κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τζομαρία Ουτζία, και η τελευταία του κυρίου Γιώργου Λάιχφριντ για την θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στου αερολιμένε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο στους εισηγητέ. Κύριε Ζασάντα, έχετε τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όδης εισηγητές για τις πολλές μακρές συνεδριάσεις μας, κατά τις οποίες μπορέσαμε να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Τώρα είμαστε λίγο πριν από την ψηφοφορία για τον κανονισμό για ε, την ε, εξυπηρέτηση. Το, η βασική ένσταση δεν είναι η απελευθέρωση του τομέα των, της ε, πηγής εξυπηρέτησης, της εξυπηρέτησης εδάφους, αλλά να προετοιμάσουμε το ευρωπαϊκό τομέα για να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όλοι θυμόμαστε πως επιστρέψαμε στις πατρίδες μας πριν από δύο χρόνια για τα Χριστούγεννα και πολλοί κολλήσαμε στα αεροδρόμια. Γιατί, Γιατί ξαφνικά ε, υπήρχε πρόβλημα με το υγρό από πάγωση των αεροσκαφών όχι επειδή το είχαν ξεχάσει να το παραγγείλουν, αλλά επειδή οι εταιρείε εξυπηρέτηση εδάφου δεν ήταν ε, προετοιμασμένε για τι καιρικέ αυτέ συνθήκε. Ω Κοινοβούλιο, προτείναμε για πρώτη φορά στην ε, ενωσιακή νομοθεσία να εισαγάγουμε ελάχιστα ε, πρότυπα ποιότητα στις υπηρεσίες εδάφους συμπεριλαμβάνοντας ε, και την ελάχιστη ποσότητα υγρού από πάγωση των αεροσκαφών για να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στο μέλλον. Όλοι μας ε, είχαμε την εμπειρία να περιμένουμε μισή ώρα και παραπάνω για να κάνουμε check-in στο αεροδρόμιο ή να περιμένουμε αρκετά λεπτά μέχρι να έρθουν οι αποσκευές αν δεν είχαν απολεστεί πριν. Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα μετά την επιβολή ελάχιστων ποιοτικών προτύπων αυτά τα προβλήματα θα μειωθούν στο ελάχιστο. Χάρη σε, αυτή, σε αυτόν τον κανονισμό έχουμε και μία έγκριση ευρωπαϊκή για τις εταιρείε εξυπηρέτησης, οπότε να μην υπάρχει πρόβλημα μια γαλλική εταιρεία να παράσχει υπηρεσίες στη Γερμανία για παράδειγμα. Τι άλλο θα αλλάξει μία διαδικασία διαγωνισμού για όλα τα αεροδρόμια για να επιλεγεί η εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους η οποία θα δραστηριοποιηθεί εκεί. Δυστυχώς η συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο το ουσιαστικό στο έγγραφο αυτό κυριαρχήθηκε από το θέμα του ανοίγματο της αγοράς στα διάφορα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Εγώ δεν το ονομάζω αυτό άνοιγμα και απελευθέρωση αλλά συνέχιση μιας πολύ ενός πολύ συντηρητικού και σόφρονος ανοίγματο της αγοράς. Γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για απελευθέρωση αυτού του τομέα αν στα μεγαλύτερα αεροδρόμια προτείνουμε μόνο να προσθέσουμε μία μόνο πρόσθετη εταιρεία εξυπηρέτησης και μάλιστα σε περίπτωση όπου το 90% των ευρωπαϊκών αεροδρομίων αυτό δεν γίνεται ούτως ή άλλως διότι δεν υπάρχουν δύο, τρεις ή τέσσερις εταιρείες αλλά υπάρχουν και οκτώ καμιά φορά. Κατά τις συζητήσεις που ακουγάτε ο εξής επιχείρημα συχνά. Θα μειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών, θα υποβαθμιστεί η ασφάλεια. Δεν αληθεύει αυτό. Μη συμπεριλάβαμε και πρόταση για ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που θα τηρούνται. Αν πέσουν κάτω από τα πρότυπα αυτά, τότε τα κράτη-μέλη μετά το, από έτοιμο από το αεροδρόμιο θα επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρείες. Θα επιβάλλουν ε, ε, ε, χρηματικό πρόστιμο. Τώρα για την επιδείνωση των συνθήκων εργασίας. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Η πρόταση της Κομισιόν συμπεριέλαβε για παράδειγμα την υποχρεωτική παράδοση των εργαζομένων στην εταιρεία που έχασε το διαγωνισμό. Τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν επιβληθεί, κατοχυρωθεί από την ε, Αρμόδια Επιτροπή. Ε, τρίτο, ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα αεροδρόμια μας. Όχι, η απελευθέρωση αυτού του τομέα έλαβε χώρα το 1996. 11 κατηγορίες ε, πήγειας εξυπηρέτησης υπάρχουν. Η αγορά για 7 έχει απελευθερωθεί πριν από 15 χρόνια και παραπάνω. Τέσσερις, ε, για τέσσερις δηλαδή υπηρεσίε αποσκευών, διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου, υπηρεσίε διαδρόμου και εφοδιασμό με κάψιμα και λιπαντικά, εκεί υπάρχει περιορισμό εισόδου στην αγορά και δεν είναι περισσότεροι από δύο οι εταιρείε. Ω ε, εισηγητή θα ήθελα να δούμε αντικειμενικά το έγγραφο αυτό. Όχι μέσα από το πρίσμα μόνο λίγων αεροδρομίων που θέλουν να διατηρήσουν το μονοπόλιο του και το μολοπόλιο για τις εταιρείες ε, ε, τις υπηρεσίες εδάφου, εδάφους, θέλουμε να δούμε τα συμφέροντα των πολλών εκατομμυρίων επιβατών που κάθε χρόνο περνούν από τα αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο κύριο Κάλλας, τους αγαπητούς συναδέλφους οι προβλέψεις μας λέγουν ότι οι αερομεταφορές μέχρι το 2030 θα διπλασιαστούν και η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη ζήτηση αυτή λόγω των περιορισμένων αερολιμενικών ικανοτήτων τις οποίες έχει. Υπάρχει ένα υψηλότατο επίπεδο ήδη στον ανταγωνισμό ανάμεσα στις διάφορες περιοχές και στις διάφορες επιχειρήσεις και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα η δραστηριότητα αυτή σε χώρες όπως ο Ειρηνικός, η Άπο Ανατολή, η νοτιο Αμερική και η Ευρώπη φαίνεται ότι χάνει μια μερίδα των αερομεταφορών λόγω και των περιορισμών των αερολιμενικών. Είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να δώσουν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις και να χρησιμοποιήσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση. Γνωρίζουμε όμως ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι διαθεσιμότητες σε επίπεδο εδαφικό, σε επίπεδο χώρου είναι περιορισμένες για νέα αεροδρόμια, για νέους διαδρόμους και γι' αυτό το θέμα της κατανομής των χρονοθυρίδων, των σλότ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Θα έλεγα ότι αυτά τα σλότς είναι κάτι που επιτρέπει στον οργανισμό να επιβιώσει τον οργανισμό των αερομεταφορών. Της 6 Νοεμβρίου έγινε δεκτή η έκθεση από την Αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου και ε, δέχεται το κείμενο του κύριου Κάλλας καταδικάζοντας βέβαια την σχέση 80% με 20%. Το κείμενο προβλέπει σαν απόλυτη καινοτομία θα έλεγα την δυνατότητα νόμιμης χρήσης των δυνατοτήτων της δευτερεύουσας αγοράς και στον τομέα των σλότ με οικονομική αποζημίωση κάτι το οποίο επιτρέπει στις αερομεταφορές να προσαρμόζουν τις χρονοτηρίδες που έχουν στη διάθεσή τους με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Αυτές οι ανταλλαγές χρονοθυρίδων θα πρέπει να γίνονται υπό την αυστηρότατη επίβλεψη των αερολιμενικών αρχών για να υπάρχει διαφάνεια και τάξη. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν στην Επιτροπή Μεταφορών θεωρήσαμε χρήσιμη τη δημοσίευση των δεδομένων για τις οικονομικές ε, έκροες από την ε, ανταλλαγή χρονοθυρίδων. Πάντα αναφερόμενοι στη δευτερεύουσα αγορά των χρονοθυρίδων ε, υπάρχουν και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες οι οποίες αποφέρουν και αυτές έσοδα που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των αερολιμενικών υποδομών. Για να υπάρξει λοιπόν μια θεμητή μορφή ανταγωνισμού ανάμεσα στους αερομεταφορείς προβλέπεται η εγγύηση της πλήρους ανεξαρτησίας του ρόλου των υπευθύνων για, τα, για τους αερολιμένες που είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας η οποία κατανέμει τις χρονοθυρίδες. Είναι υπεύθυνη για την κατανομή των χρονοθυρίδων με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή. Πρέπει λοιπόν να έχουν πλήρη ανεξαρτησία και σε επίπεδο οικονομικό πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να είναι ανεξάρτητες από τις αεροπορικές εταιρείες και σε επίπεδο λειτουργικό. Και ταυτόχρονα οι αρχές αυτές πρέπει να συντάσσουν μια ετήσια έκθεση που να περιγράφουν την ετήσια κίνηση και αλλαγή στην αγορά των χρονοθυρίδων. Υπάρχει και το θέμα του επιβολής κυρώσεων, το οποίο βέβαια εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να σέβεται συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες πλευρές, τις οποίες θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Αναφέρομαι σε κάποιες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί πρώτον στην επανένταξη της ε, αλληλοδιαδοχής η οποία προβλέπεται στο αρχικό κείμενο και δεύτερον να υπάρξει ένας νομικός ορισμός των χρονοθυρίδων, κάτι το οποίο να εξηγεί δηλαδή με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ενοικίαση σλότς ε, δηλαδή και αερολιμενικές αρχές, πολίτες ε, ε, ανεξάρτητοι και φυσικά αεροπορικές εταιρείες. Αυτά θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους, Λίχτενμπεργκερ, Σασόλη, Ρούτσεκ και άλλους γενικά, οι οποίοι προσπάθησαν και έχουν συνεισφέρει τα μάλα στη σωστή παρουσίαση του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το σημείο κινήσεως για την έκθεση αυτή είναι σε γενικές γραμμές το ακόλουθο. Υπήρχε η πονία ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέτρα κατά της συγχωρήπανσης από τα αεροσκάφη είναι ακατάλληλα και ασυντόνιστα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να υποβάλει πρόταση νομοθετική που θα άλλαζε την κατάσταση με την έννοια ότι θα αποκατασταθεί μια ενιαία προσέγγιση και ότι εκείνη που ε, πρέπει να... Ε, εκείνη που πρέπει να λάβουν υπόψη την οδηγία, να έχουν μια προστασία. Είτε είναι κάτοικοι που μένουν κοντά, είτε χρησιμοποιούν τα ε, αεροδρόμια και τα αεροσκάφη. Νομίζω ότι είναι σχετικά ε, λογικό αυτό. Επίσης, ε, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα προβλήματα με την ηχορύπανση, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, οξύνονται όλο και περισσότερο και γι' αυτό έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει. Ένα πράγμα όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να το κάνει η έκθεση αυτή. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε ανώτατα όρια θορύβου, ούτε μπορούμε να ρυθμίσουμε τι είναι αποδεκτό σε επίπεδο θορύβου στην Ευρώπη και τι όχι. Θα ρυθμίσουμε μόνο το πώς θα υπάρξουν μέτρα προς, η προστασίας από το θόρυβο και αυτό ανταποκρίνεται και στην προσέγγιση του ΙΚΑΟ που λέει ότι πρώτα θα πρέπει να ληφθούν οι ποιότερα μέτρα και αν δεν έχουν αποτέλεσμα ούτε αποτελεσματικά ούτε αποδοτικά τότε θα ε, κλιμακωθούν τα μέτρα μέχρι την απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων. Το πρόβλημα λεπτομερέστερα που μας απασχολεί ως επιτοπλίστων εδώ είναι τριπλό. Πρώτο, πώς τα αεροσκάφη τα οποία οριακά συμμορφούνται προς τις διατάξεις, σταδιακά θα αποσυρθούν. Νομίζω ότι εδώ βρέθηκε μια καλή λύση, δηλαδή με μια μεταβατική περίοδο και σταδιακά να αποσυρθούν αυτά τα θορυβόδη, να αντικατασταθούν από λιγότερο θορυβόδη. Αυτό ήταν σωστό. Το δεύτερο ζήτημα, τι γίνεται με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως νομοθέτη. Εδώ δεν συμφωνήσαμε απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά που αποφασίσαμε στην Επιτροπή και αυτά που θα αποφασίσουμε μάλλον και στην Ολομέλεια είναι ότι όταν είναι πολιτικά τα θέματα που πρέπει να αποφασιστούν τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των ε, πολιτών θα πρέπει να αποφασίσει και όχι η Κομισιόν με κατεξουσιοδότηση πράξη. Όταν όμως πρόκειται για τη λήψη τεχνικής φύσεως αποφάσεων, τότε μπορεί να ε, ε, το κάνει η Κομισιόν με κατεξουσιοδότηση πράξη. Το τρίτο και δυσκολότερο πρόβλημα ήταν το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική πρόταση προέβλεπε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να έρει και τα εθνικά μέτρα προστασίας από το θόρυβο. Λάθος αυτό. Νομίζω ότι κάθε ομόσπονδο κρατήδιο ε, μπορεί κάλλιστα από μόνο του πιστεύω να κρίνει αν ένα μέτρο προστασίας από το θόρυβο χρειάζεται και σε ποιο βαθμό χρειάζεται. Και νομίζω ότι οι δυνατότητες που είχε μέχρι τώρα η Κομισιόν μέχρι τη διαδικασία ε, επιπαραβάση κατά των κρατών μελών ε, ήταν επαρκέ για να προστατεύεται το ενωσιακό ε, δίκαιο. Φροντίσαμε επίσης στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνεται καλύτερα, να συνεργάζεται καλύτερα με τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, ούτω ώστε να βελτιωθεί το συνολικότερο επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κάνω και μια προσωπική παρατήρηση, τελείωσα κατά τα άλλα. Όταν ανέλαβα την έκθεση σκέφτηκα καταρχήν ότι είναι ανεπίλητο το πρόβλημα. Όμως είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με συναδέλφους οι οποίοι ε, έδειξαν ιδιαίτερη ε, αφοσίωση και δέσμευση. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους θερμά και ευχαριστώ ιδιαίτερα του υπεύθυνου συνεργάτες μου, αρμόδιου, ε, για το φάκελο αυτό στο γραφείο μου. Γιατί χωρίς την εξαιρετική του εργασία δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι συνάδελφοι. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Κάλλας να μας παρουσιάσει την άποψη της Κομισιόν. Πρόεδρε, εξότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να υπενθυμίσω για ποιο λόγο ε, παρουσίασε η πρόταση, την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι το Δεκέμβριο για τα αεροδρόμια. Όπως μας είπαν ε, όλοι οι συγητές, ε, είναι εύκολο να οικοδομήσουμε νέους διαδρόμους, να διευρύνουμε τα αεροδρόμια σήμερα στην Ένωση. Ταυτόχρονα όμως ε, είναι κορεσμένος ο ευρωπαϊκός ε, χώρος ε, και αυτό συμμεπάγεται καθυστερήσεις για το ίμιση το σύνολο των πτήσεων σε ολόκληρο το δίκτυο μέχρι το 2030. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε μετριοπαθείς αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία ως προς τις υπηρεσίες εδάφους των αεροδρομίων για να βελτιώσουμε τη δυναμικότητα των αεροδρομίων. Ας αρχίσω με τις υπηρεσίες εδάφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζασάντα, ε, ε, τον εισηγητή μας ε, για τη δουλειά που έκανε τους περασμένους μήνες γιατί πραγματικά δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ε, πάντως είναι ισοσκελισμένη η πρότασή μας. Ε, ε, καλύπτουμε την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υψηλότερη ποιότητα στου αερολιμένε της Ένωση, ε, προαγάγοντα ε, και την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν προτείνουμε την άγρια απελευθέρωση. δηλαδή το να περάσουμε από την σημερινή κατάσταση, δηλαδή δύο παρόχους στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης σε τρεις για μια περιορισμένη κατηγορία υπηρεσιών σίγουρα δεν συνιστά άγρια απελευθέρωση. Ε, και προτείναμε διάφορα μέτρα για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και να κατοχυρώσουμε την καλή ποιότητα. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι διακυβεύεται η ασφάλεια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση περάσει από το σύστημα των δύο παρόχων στο σύστημα των τριών. Δεν ευσταθεί αυτό ήδη. Έχουμε στην πλειοψηφία των κρατών μελών μια κατάσταση όπου επιτρέπονται οι τρει επάροχοι και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ασφάλεια. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξαναλέω, είναι ένα μετριοπαθέ βήμα προς άνοιγμα τη αγορά, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε ε, την κοινωνική ισότητα και ενισχύουμε τα πρότυπα. Με το 2007 θα ήθελα να σα υπενθυμίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του ψηφίσματο τη Αν Γένσεν απίφθινε έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την ε, κατάσταση για τι υπηρεσίε εδάφου. Μέσα σε αυτό το ψήφισμα ζητήσαμε αύξηση του ελαχίστου αριθμού παρόχων και ζήτησε δράση επί τη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Απαντήσαμε λοιπόν με αυτή την εξισορροπημένη πρόταση που ε, προφανέστατα επιδέχεται βελτιώσει, αλλά θα πρέπει να δράξουμε με την ευκαιρία. Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα των χρονοθυρίδων τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Ουτζία για τη δουλειά που έκανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ω επιτοπλίστων τι τροπολογίε που κατέθεσε η Επιτροπή Μεταφορών. Εν συντομία, θα ήθελα να τονίσω κάποια σημεία κεφαλαιόδου σημασία. Σε πρώτον, ε, δευτερογενή εμπορία. Ε, οι μηχανισμοί τη αγορά μπορούν να μα βοηθήσουν ε, για να εξασφαλίσουμε ότι οι χρονοθυρίδε, ε, που είναι περατό πόρο, θα χρησιμοποιούνται καλύτερα από του αερομεταφορεί που είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των χρονοθυρίδων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι περιφερειακέ εναέρειε διασύνδεσει θα προστατευτούν πλήρω. Αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο των τροπολογιών Λοιπόν για τις πιθανέ επιπτώσεις για τέτοιου είδου διαδρομές στη δευτερογενή αγορά. Οι συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά πρέπει να συνοδεύονται από ποιοτικά κριτήρια. Η διαδικασία χορήγηση των χρονοθυρίδων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως... Ε, μία τροχοπέδη, ένα, εναντίον της ε, ε, λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς. Για το θόρυβο θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών και τον κύριο Γιώργο Λάιχφρυντ, τον εισηγητή της, για όλα αυτά που έκανε για να επεξεργαστεί την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπόρεσε ο εισηγητή ε, να τροφοδοτήσει μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Ε, το πρόβλημα του θορύβου δημιουργεί πίεση σε περιφερειακό πολιτικό επίπεδο. Οποιαδήποτε όμω προσπάθεια μετριασμού του θορύβου επηρεάζει ολόκληρη τη βιομηχανία. Και αυτή είναι η καρδιά του προβλήματο. Η χορύπανση των αεροδρομίων είναι ένα τοπικό πρόβλημα, ενώ επηρεάζεται όλη η βιομηχανία για τα μέτρα, από τα μέτρα συγγνώμη, που χρησιμοποιούμε για τον μετριασμό του θορύβου θορύβου. Το προτινόμενο δικαίωμα ελέγχου από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μα βοηθήσει ε, ούτω ώστε να επιτύχουμε την επιθυμητή ισορροπία στην πράξη. Τέλος, Πάλι για το κομμάτι του θορύβου του πακέτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί την, ε, την ε, εισαγωγή ε, του ορισμού των αεροσκαφών που οριακά συμμορφούνται με τα πρότυπα, διότι δεν έγινε εμπρόθεσμα. Αυτά τα αεροσκάφη είναι τα πλέον θορυβόδη στο στόλο και επιφέρουν ένα δυσανάλογα μεγάλο άχθος ως προς το, την χορύπανση. Γι' αυτό και με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου οι εθνικές αρχές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα αποτελεσματικά ως προς το κόστος. Ε, προσβλέπω στην ενδιαφέρουσα συζήτηση και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a parlament szakbizottságainak a véleményét ismerhetjük meg. Elsőként a foglalkoztatási... Πρώτος ομιλητής εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης είναι ο κύριος Μάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. χιλιάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν σήμερα, εργαζόμενοι στα αεροδρόμια. Και εδώ, πριν από το, έξω από το Κοινοβούλιο, όπως και στις Βρυξέλλες, σχετικά με τα σχέδια περαιτέρω ανοίγματο τη αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μήνυμα τη Επιτροπή Μεταφορών δεν το έλαβε υπόψη και δεν απέσυρε την πρότασή τη. Τη θέση τη Επιτροπή ε, Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων την αγνώρισε επίση. Στην έκθεσή μου, οι θέσει εργασία ε, πρέπει να ε, διασφαλίζονται. Ε, μια ριζική, ένα ριζικό άνοιγμα της αγοράς οξύνει τα προβλήματα. Ε, οι συμβάσεις αορίστου χρόνου μειώνονται, το μισθολογικό ντάμπινγκ απειλεί. Ε, χρειάζεται καλό σύστημα εξυπηρέτησης εδάφους από καταρτισμένο προσωπικό με, όχι με εμβαλωματικές λύσεις και σεμινάρια. τα κοινωνικά θέματα ε, έχουν αποφασιστεί από, στο σχετικό κανονισμό από, το προ, από το, την πρόταση ε, της ε, Κομισιόν καταφέραμε να ε, βγάλουμε τα, κάποια δικαιώματα για, κοινωνικά για τους εργαζομένους. Ε, επίσης ε, αναφέρεται ε, εγγύηση της θέσης εργασίας όταν κλείνουν κάποιες εταιρείες. Επίσης στον τομέα της εκπαίδευσης κατάρτισης στο άρθρο 34 υπάρχει ε, μια προστασία απέναντι ε, σε αυτήν την, ε, την ακραία απελευθέρωση. Το σχέδιο Β είναι η πρόταση της Επιτροπής Απασχόλησης. Λοιπόν, η Ευρώπη χρειάζεται κοινωνικό πρόσωπο. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα για καλή αμοιβή και επιτέλους για κοινωνική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ε, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγιάλα Σέντερ. Εκπροσωπώ λοιπόν την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εμείς εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη στα πλαίσια της ε, νομοδότησης αυτής οι απόψεις ε, γενικά των ε, εκπροσώπων των τοπικών αρχών στον τομέα της τεχνικής συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο θα μας επέτρεπε να έχουμε μια πληρέστερη αντίληψη για τα πράγματα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις εκπομπές ε, καυσαερίων. Εμείς είχαμε ζητήσει επίσης να υπάρξουν διαβουλεύσεις όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο των κοινοτήτων οι οποίες θίγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις εμπειρίες που θα μας επέτρεπε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν με μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά μπορούν να γίνουν αντιληπτά και με γενικότερο πιο σφαιρικό τρόπο. Έτσι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αποτελεσματικά το θέμα των αεροδιαδρόμων, ε, ακούγοντας προσεκτικά, εν πάση περιπτώσει, την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί ένα κοινωνικό πακέτο, ένα κοινωνικό πακέτο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν έγινε δεκτό. Ευχαριστώ από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών, η κυρία Γκαλσπέλς, δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Ζάσαντα, ο συνεισηγητής, παρουσίασε ένα διτό πρόβλημα. Οι υπηρεσίες εδάφους δεν είναι παρκώς αποτελεσματικές και η ποιότητα δεν καλύπτει ε, τις αξιώσεις των χρηστών. Πρότεινα μέτρα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εδάφους και ενίσχυση της ε, ε, αποτελεσματικής λειτουργίας ε, των αερολιμένων. Η πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών συνιστά πρόοδο από νομοθετικής πλευράς, όμως εκκρεμούν ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και να τα επεξεργαστούμε. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ενίας Αγοράς, κρίνουμε ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι αναγκαίο το άνοιγμα της Ενίας αγοράς, διότι την παρούσα στιγμή θα συνεπάγεται αυτό αυξημένη πίεση ε, για τους αερομεταφορείς και τους παρόχους των υπηρεσιών. Προτείνουμε λοιπόν για τους αερολιμένους που είχαν τζίρο τα τελευταία τρία χρόνια ε, τέτοιο που να καλύπτουν 5 εκατομμύρια επιβάτες ε, να χρησιμοποιηθούν ως όριο ε, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται μια σύσταση προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές ε, που θα γνωμοδοτούν αν θα κρίνουν δηλαδή απαραίτητη αύξηση του αριθμού ε, των παρόχων υπηρεσιών λόγω περιφερειακών ή τοπικών αναγκών του συγκεκριμένου αερολιμένα. Ε, πιστεύω ότι αν δεν προσέξουμε θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε εύκολα σε μείωση των ε, μισθών, σε δημιουργία επισφαλών θέσεων απασχόλησης, σε ε, επιδείνωση των κανόνων για τις ε, θέσεις εμερικής απασχόλησης ή για την εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού. Αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος και τώρα... Εξ ονόματος ε, των πολιτικών ομάδων ε, θα ακούσουμε τους ομιλητές Κάρλο Φιντάντσα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ούτζιας ε, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε σχετικά με την ε, ε, χορήγηση των χρονοθυρίδων. Είχαμε κάποια προβλήματα με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταφέραμε να επιφέρουμε τροποποιήσει στην Επιτροπή, επιτυγχάνοντα μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προ τη χρήση των χρονοθυρίδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΛΚ υποστήριξε εξ αρχή τη διατήρηση του κανόνα 80-20 ε, σε σχέση με του κανόνε χορήγηση και κατανομή των χρονοθυρίδων, ε, ούτω ώστε να μην πλήξουμε την ισορροπία ενό συστήματο που λειτουργεί ε, αισίω και για να μην δημιουργήσουμε στις δυσκολίες στην αγορά. Το θέμα των ακυρώσεων είναι κάτι που πρέπει να δούμε, όπως επίσης και το θέμα της επιβολής κυρώσεων σε ανάρμοστες συμπεριφορές. Θα πρέπει οι κανόνες να είναι διαφανέστεροι, να υπάρξουν έλεγχοι και για τη δευτερογενή αγορά, έτσι ώστε να αποφύγουμε καταχρήσεις από πλευράς των αερομεταφορέων. Για πρώτη φορά έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τις υποδομές της αερολιμανικές οι οποίες ε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της φορητικότητας. Ε, εδώ υπάρχει και το θέμα των υπηρεσιών εδάφους. Εγώ θέλω να στηρίξω εδώ στην εργασία του εισηγητή του κυρίου Ζασάντα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να παραπεμφθεί προς ε, νέα εξέταση ε, η πρόταση, όχι ότι δεν έχει γίνει καλή δουλειά μέχρι τώρα, έχουν υπάρξει σημαντικά βήματα και στον τομέα τον κοινωνικό με τις προσπάθειες και τη συνεισφορά της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Εμείς ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δεχθούμε την πρόταση αυτή εξετάζοντάς τις πάρα πολύ προσεκτικά όμως. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλιστών, ο κύριος ε, Σαϊνταλ Αλκαντράουι. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συζητητές και τους σκιώδεις συζητητέ για το έργο τους. Ήταν πολύ εξαιρετικό. Ακόμη όμως έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Είναι πολλές οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί και εμείς ως ομάδα διαφοροποιούμεθα από άλλους. Ο κύριος Λάιχτφριντ βρήκε καλή ισορροπία για το θόρυβο και την εναρμόνιση στην νομοθεσία για να αποφεύγεται η χορύπανση. Υπάρχουν καλές προτάσεις από την άλλη πλευρά. Η αρχή της επικουρικότητας για να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα πολύ λεπτών διαπραγματεύσεων ε, και μηχανισμών που έχουν εγκριθεί για την ελαχιστοποίηση της κατανομής ε, και την ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών να υπάρχουν οι δυνατότητες επανεπένδυσης κεφαλαίων εκεί. Θέλουμε όμως ως ομάδα να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο από αυτά. Θέλουμε να είναι πιο ευέλικτο το σύστημα με τις ε, ε, σειρές των χρονοθυρίδων να είναι πιο ευέλικτο. Πάντως πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Και η, περαιτέρω απελευθέρωση του συστήματος ε, εξυπηρέτησης δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Δηλαδή δεν συμφωνούμε ούτε με τον εισηγητή ούτε με την Κομισιόν εδώ. Νομίζω ότι ε, επιμένουμε πολύ στην μείωση, το, μειωμένη παροχή υπηρεσιών και την αύξηση του αριθμού των εταιριών που πρέπει να συμμετέχουν. Εμείς δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει να ε, το δούμε έτσι. Ε, το ζήτημα είναι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, γιατί ορισμένοι, καμιά φορά είναι μικρότερο το αεροδρόμιο και έχει μικρές εταιρείες που δουλεύουν καλά τα κράτη-μέλη λοιπόν που θα πρέπει να αποφασίσουν ε, για το ζήτημα αυτό και θα ζητήσουμε να ε, το απορρίψουμε αυτό. Πάντως είμαστε διαθέσιμοι για να διαπραγματευτούμε. Εάν υπάρξει κάποιο ε, άνοιγμα προς την κατεύθυνση των προτάσεών μας πιστεύουμε ότι οι σημερινοί κανόνες δεν είναι καλοί ούτε αυτοί. Αλλά νομίζω ότι αυτά που θα προταθούν σήμερα είναι ανεπαρκή και θα ψηφίσουμε κατά. Ευχαριστώ πολύ εξ ονόματο τη ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, ο κύριος Βολφ Κλίντς. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, τα κράτη-μέλη ήδη από σήμερα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τα ίδια σε ποιο βαθμό θα απελευθερώσουν τις υπηρεσιες εδάφου. εδάφους. Πολλά κράτη-μέλη το αξιοποίησαν αυτό σε μεγάλο βαθμό, άλλες σε λιγότερο βαθμό και υπάρχει βέβαια και διαφορά σε σχέση με τα αεροδρόμια και το μεγεθό του. Η Κομισιόν τώρα θέλει να μειώσει λίγο αυτή, αυτή τη διαφορά στα αεροδρόμια και ελπίζει ότι με την αύξηση του ανταγωνισμού θα βελτιωθεί και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Ως εδώ καλά. Μάλιστα η Κομισιόν θέλει και ε, ριζική απελευθέρωση. Εγώ ως φιλελεύθερος είμαι καταρχήν υπέρ της απελευθέρωσης, ε, αλλά μόνο όταν επιτυγχάνεται ο καθαυτός στόχος μας. Εκεί έχω πρόβλημα. Εξίδια πείρα ξέρω ότι δεν είναι ο αριθμός των υπηρεσιών που κρίνει το καλό σερβις, την καλή ποιότητα, αλλά το πώς οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες εδάφους είναι εξειδικευμένοι, Ποιε είναι οι συνθήκε εργασία και πόσο ενδιαφέρονται για τη δουλειά του. Εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι δηλαδή με τυφλή αύξηση των ε, υπηρεσιών που συμμετέχουν στην εξυπηρέτηση θα επιτύχουμε το στόχο. Αυτό το βλέπουμε κριτικό πνεύμα. Ε, είμαι, θα προτιμούσα πιο περιορισμένη απελευθέρωση όπως την προτείνει η Κομισιόν, πάντα με την προϋπόθεση ότι τα κράτη-μέλη σε τελευταία ανάλυση θα αποφασίζουν ε, γνωρίζοντας ε, τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο. Είναι μεγάλες οι διαφορές μεταξύ αεροδρομίων, το ξέρω. Το, το δικό μου αεροδρόμιο είναι το, το Φραγκφούρτη, είναι της Φραγκφούρτης και τώρα ε, ε, με την ε, διεύρυνση του οδικού δικτύου έχει μειωθεί ο διαθέσιμος χώρος για το αεροδρόμιο. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ναι, με, την, με μέτρο απελευθέρωση και πάντοτε θα πρέπει να έχουν λόγο τα κράτη-μέλη εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Egy με Μία μπλε κάρτα βλέπω. Ο κύριος Φαντάλεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι δεν κατανοώ, κατανοώ αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Κλίντς. Ο κύριος Κλίντς είναι υποτίθεται φιλελεύθερος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσει περισσότερες δυνατότητες στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αυτά τα οποία λέγει ο κύριος Κλίντς δεν θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε στο επίπεδο φιλελευθεροποίησης το οποίο θα προτιμούσαμε. Αυτό το οποίο ζητάει ο κύριος Κλίντς το κάνει η Επιτροπή ε, Απασχόλησης με τον πολιτισμένο και κατάλληλο τρόπο μας οδηγεί στη φιλελευθεροποίηση του τομέα χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί είστε κατά. Ε, δεν κάνω πολεμική. Αυτό που λέω είναι ότι το στόχο της απελευθέρωσης θα πρέπει να τον προσεγγίσουμε με μέτρο. Οι ιδιαιτερότητες ενό τοπικού αεροδρομίου πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη. Δεν είναι όλα τα αεροδρόμια ίδια. Ε, σκεφτείτε τη Φραγκφούρτη. Εκεί έχουμε μεγαλύτερη μεταφορική δυνατότητα, ε, αλλά το Terminal 3 που ε, θα έπρεπε να απορροφήσει την ε, ε, πρόσθετη χωρητικότητα ακόμη δεν έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι εδώ θα απελευθερώσω, θα διπλασιάσω τον αριθμό των υπηρεσιών εδάφους. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει κάτι τέτοιο με αυτή τη σειρά. Γι' αυτό λέω με μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές συνθήκες εργασίας, την εξειδίκευση, ούτως ώστε το σέρβις και η ποιότητα να είναι εγγυημένες. Ο κύριος Ζασάντα τώρα θα πάρει το λόγο. Ε, ε, έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Κλίνς και εγώ. Τι εννοείται μιλώντας ε, για σπαστική, άγρια απελευθέρωση, τι εννοείται. Από ό,τι κατάλαβα, ε, εσείς γνωρίζετε η κατάσταση για το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και αληθεύει ότι έχουμε δύο παρόχους. Ο ένας ε, καλύπτει το 85% των υπηρεσιών και ο δεύτερος το 15%. Λοιπόν, στην τροπολογία μου εγώ εισηγήθηκα τρεις. Αύξηση από δύο σε τρεις παρόχους. Ε, δεν αυξάνουμε κατά 100% αλλά κατά 50%. Ως προς τα κοινωνικά ζητήματα... Νομίζω ότι όλοι ζήσαμε τις χιλιάδες των συνδικαλιστών που ε, ε, διαδήλωσαν μπροστά στο, στο κοινοβούλιο και ξέρετε τι μου είπαν. Μου είπαν πω θέλουν να αναπαιμφθεί στην Επιτροπή Μεταφορών το κείμενο. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Πρόεδρο, με την μπλε κάρτα έχετε στη διάθεσή σας, κύριε Κλίντ, σε μισό λεπτό για να απαντήσετε. Δεν θα πω πολλά μετά την παρέμβαση του κυρίου Σασάντα, δεν είναι ερώτηση, μάλλον σχόλιο έκανε. Νομίζω ότι καλά θα κάναμε να αφήναμε τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν με τους δικούς τους νόμους, την νομοθεσία τους και να ανταποκριθούν στα προβλήματα. Επαναλαμβάνω μόνο αυτό που είπα, στο βαθμό που οι τοπικές ε, συνθήκες ε, είναι ε, συγκεκριμένες και δεν επιτρέπουν την αύξηση των ε, παρόχων υπηρεσιών εδάφους, δεν πρέπει ούτε εμείς να το σκεφτόμαστε. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν πότε θα έρθει η ώρα να προχωρήσουν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η δική μου θέση. Φαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, έχουν έρθει τα πράγματα, έχουν γυρίσει τα πάνω κάτω. Έχουμε προβλήματα στη Φραγκφούρτη, το καταλαβαίνω. Και εδώ έχουμε τον φιλελεύθερο κύριο Κλίντς, ο οποίος προσπαθεί να παρεμποδίσει την εξέλιξη της αγορά αυτής στην Ευρώπη, μια κλειστή αγορά, η οποία θα πρέπει να γίνει δεκτική και πολύ πιο ανεκτική. Δεν καταλαβαίνω, έπρεπε να λειτουργήσετε με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να καταθέσετε τροπολογίες, να αναφερθείτε στον κατώτερο μισθό στην Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει θα είχαμε λάβει με διαφορετικό τρόπο υπόψη την άποψή σας. Τώρα αυτό το οποίο λέτε δεν έχει ε, θέση. Παρακαλώ απαντήστε κύριε Κλίντ σύντομα. Δεν σας καταλαβαίνω συνάδελφε. Ε, ε, δεν είπα εγώ ότι θα πρέπει ε, να ε, μιμηθούν τη Φραγκφούρτη όλοι. Ε, τα κράτη-μέλη είπα ότι πρέπει να κρίνουν τα αεροδρόμια τους με βάση τις τοπικές συνθήκες. Αν πούν κάποιοι ότι είμαστε εξοπλισμένοι έτσι και έχουμε υποδομή για να διπλασιάσουμε τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εδάφους, κανένα πρόβλημα, δεν θα τους σταθώ εμπόδια εγώ. Κάλερ και ε, στη συνέχεια δεν θα ακούσουμε άλλες ερωτήσεις με την μπλε κάρτα. Κύριε Βαντάλεν, γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μπορούν να απελευθερωθούν τα πάντα. Όχι, παρέμβαση του Προέδρου. Με συγχωρείτε κύριε Γκάλερ, η μπλε κάρτα αφορά μόνο τον ε, ομιλητή δεν μπορεί να έχετε μπλε κάρτα για να απευθυνθείτε σε άλλον συνάδελφο που έκανε ερώτηση με μπλε κάρτα. Αυτή ο κανονισμός. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και για την ετοιμότητα του αγορητή που έδωσε τις απαντήσεις του. Και τώρα θα συνεχίσουμε. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ Εύα για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ συνάδελφοι υποβέλτιστη η πρόταση, οπότε δύσκολα να δώσει κάτι καλό. Ευχαριστώ τους εισηγητές που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν πάντως. Τώρα για τις υπηρεσίες εδάφους. Η πρόταση απερίφθη στην Επιτροπή ε, διότι λίγα θετικά αναμένεται να δώσει κοινωνικό ντάμπινγκ στα αεροδρόμια, χειρότερε συνθήκε αμοιβή και απασχόληση, λιγότερη κατάρτιση και όλα αυτά γιατί υπόσχονται μείωση του κόστου που ε, συνήθως μετακυλίεται και στους επιβάτες. Ένα ε, περαιτέρω βήμα απελευθέρωσης είναι, θεωρούμε, τελείως περιττό. Αυτό που με ενόχλησε ήταν ότι η Κομισιόν έκανε έντονο lobbying μετά την απόφαση της Επιτροπής για να περάσει παρόλα αυτά η πρότασή της. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, σεβαστούμε μια ηλυμένη απόφαση. Ε, ε, υπάρχουν εδώ και οι μάρτυρες οι συνάδελφοι. Τώρα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας έδειξε πόσο ε, βλαβερή είναι η χορύπανση την ημέρα αλλά και τη νύχτα. Ο θόρυβος ευθύνεται για προβλήματα υγείας και για μεγάλη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στους κατοίκους κοντά στα αεροδρόμια αντί να προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες για τους ε, κατοίκους κοντά στα αεροδρόμια και να προωθήσουμε τις ε, ε, καινοτομίες, η Κομισιόν τι κάνει, ένα πράγμα μόνο. Θέλει να περιορίσει τις περιφερειακές πτήσεις αν κάποιος ανταγωνιστής βλέπει οικονομικό μειονέκτημα. Αυτό ως προσέγγιση είναι εντελώς λάθος από την αρχή. Χειρότερο δεν μπορεί να παρουσιαστεί το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες ε, αν δεν ε, απαλληφθεί το σχετικό εδάφιο που θα το καταψηφίσουμε. Γιατί ήδη δυσκολεύονται πολύ οι κάτοικοι κοντά στα αεροδρόμια να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα όταν είναι αυξημένη η κυκλοφορία. Και η πρόταση αυτή, η δική σας κύριε Επίτροπε, ε, θεωρώ ότι δεν είναι ε, καλά μελετημένη ή είναι πολύ μονόπλευρη και ε, λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των λόμπι των αεροδρομίων. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Φαντάλεν θέλει να σας υποβάλει μια ερώτηση. Δέχεστε να απαντήσετε, κυρία Λίχτενμπέργκερ, ναι? Ωραία. Φαντάλεν, μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι δύσκολη συζήτηση, αλλά άκουσα προσεκτικά την παρέμβαση της κυρίας Λίχτεμπεργκερ που λέει ότι με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί δεν πρόκειται να έχουμε μια ευτική κατάληξη. Πράγματι το σύστημα το οποίο έχουμε στην Ευρώπη δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Αυτό προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε. Α κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην Επιτροπή Μεταφορών για να ξεφύγουμε από αυτή την κακή κατάσταση και να βρούμε μια κάποια λύση. <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση βέβαια δεν άκουσα, αλλά τι θέλετε το ποιο πακέτο για τα αεροδρόμια θέλετε να πάει πίσω στην Επιτροπή ή τι. Δεν, δεν με ρωτήσατε κάτι. Γι' αυτό τι να σας απαντήσω. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Αυτός ο αποκλειστικός προσανατολισμός προς το οικονομικό όφελος και την ε, μεγάλη απελευθέρωση τον θεωρώ λάθος. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Και δεν είναι εξισορροπημένη πρόταση και γι' αυτό τη θεωρώ αδύναμη πρόταση. Κυρία Πέλς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ζητήσω από τον Πρόεδρο να μην συνεχίσει αυτή τη διαδικασία των μπλε καρτών γιατί νομίζω ότι όλα αυτά ε, θα έπρεπε να είχαν λεχθεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και τώρα δεν μας ε, βοηθούν να προχωρήσουμε. Ε, με επικρίνεται όμως βλέπω ότι πολλοί διαφωνούν μαζί σας Uh, Διαδικαστικά, για να απαντήσω στην κυρία συνάδελφε, εγώ ήμουν σκιώδης ε, πάνω στο θέμα αυτό της, ε, ε, των υπηρεσιών εδάφους και δεν έκανε τίποτε για να ε, εμποδίσω τη συζήτηση. Ε, δεν μπορείτε να λέτε ότι ε, τα είπαμε στην Επιτροπή. Είναι δημοκρατικό μου δικαίωμα να κάνω ερωτήσεις στην Ολομέλεια όπως έκανα και στην, στη συνεδριάση της Επιτροπής. Δεν μπορείτε να το εμποδίσετε αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Και ο πρόεδρος έχει τη διακριτική ευκαιρία να δεχτεί ή να μην δεχτεί την μπλε κάρτα. Προχωρούμε τώρα στη γνώμη των Ευρωπαίων Συντηρητικών, η Ζακλίν Φωστέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάει πολωνικά η κυρία Φώστερ. Κάνατε μια εξαιρετική δουλειά. Θα ήθελα να μιλήσω για τις υπηρεσίες εδάφους. Οι συντηρητικοί Βρετανοί έχουν υποστηρίξει ιστορικά θα έλεγα την απελευθέρωση. Οι εμπειρίες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι επιτυχής. Θα πρέπει να ανοίξουμε στον ανταγωνισμό. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα τα οποία επηρεάζουν ορισμένους συναδέλφους εδώ και χώρες. Αλλά για αυτούς τους λόγους ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μην υποστηρίξουμε τη συγκεκριμένη έκθεση. Καταρχάς τα υψηλά επίπεδα ε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβάλλονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Απαιτούνται ε, ελάχιστα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και βασική προϋπόθεση είναι να μην αυξάνεται το κόστος το οποίο υφίστανται οι αερομεταφορείς. Όταν ένας εργολάβος, σαν παράδειγμα, αντικαθιστά μία επιχείρηση, απαιτείται να προσλάβει πολλές φορές το προσωπικό της προηγούμενης επιχείρησης, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα συνεχίζω να ομιλώ ως εκπρόσωπος των συντηρητικών, των Βρετανών συντηρητικών, για τις χρονοθυρίδες. Θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολη. Ζήτησα επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι αλλαγές μπορεί να γίνουν υπό την υφιστάμενη νομοθεσία δεν μου έχει δώσει απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι βλέπουμε την έλλειψη ε, χωρητικότητας, ε, αλλά ξέρουμε ότι για να λύσουμε το θέμα πρέπει να δημιουργήσουμε νέους διαδρόμους στα αεροδρόμια. Εμείς έχουμε ακολουθήσει μια τέτοια πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο που εν μέρει έχει καλύψει τις ανάγκες μας. Εμείς δεν θα πρέπει τα έσοδα από την χορήγηση αυτών των χρονοθυρίδων να δίδονται χωρίς έλεγχο στην κυβέρνηση αλλά σε αυτούς οι οποίοι βελτιώνουν τις υποδομές. Το θέμα του συντονισμού της κατανομής των χρονοθυρίδων είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να ε, προχωρήσει με την καλύτερη δυνατή μορφή συντονισμού. Έχω τρία λεπτά λέει η κυρία Φώστερ και συνεχίζει. Το 80 και 20 είναι κάτι το οποίο βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Πιστεύω επίσης ότι το θέμα των χρονοτηρίδων αν το αφήσουμε ως έχει θα ήταν προτιμότερο. Το θέμα του θορύβου τώρα, ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στον τομέα θα έλεγα της, της It's important to point out that all European... το θέμα, είναι θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της επικουρικότητας. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αντιμετώπιση του. Το θέμα ε, εδώ του ορισμού και των κατηγοριών των αεροσκαφών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Ξοδέψαμε 9 μήνες εν πάση περιπτώσει σε αυτό το πακέτο και ε, πολλοί διαφωνούν με τα συμπεράσματα για διαφορετικούς ενταλώς λόγους. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει ε, να παραδεχθούμε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην παγιδευτούμε μόνοι μας ε, στους κανόνες μας και θα πρέπει να διευκρινίσουμε με σωστό τρόπο πώς θα διευκολύνουμε αυτούς που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς. Η κυρία Φώστερ λοιπόν τελείωσε. Συγγνώμη που σας διάκοψα, λέει ο πρόεδρος αλλά δυστυχώς μου είχαν πει στον κατάλογό μου ότι είχατε 1,5 λεπτό. Γι' αυτό στάθηκα γενναιόδωρο απέναντί σα και σας άφησα να ξεπεράσετε τα τρία λεπτά. Ζητώ συγγνώμη όμως που σας διάκοψα. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Βίλς. 1,5 λεπτό σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η Επιτροπή Μεταφορών, την πρόταση της Κομισιόν ήδη πολλές φορές και κατα... Ε, ήδη κατά πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση για τις υπηρεσίε εδάφους. Ε, θα ήθελα αύριο να ε, απορρίψουμε επίσης την πρόταση ακολουθήστε την ψήφο της αρμόδιας επιτροπής. Η έγκριση της πρότασης θα συνιστούσε μισθολογικό ντάμπινγκ και θα άνοιγε τις πύλες διάπλατα στα αεροδρόμια γι' αυτό. Επίσης δεν θα πρέπει να αμοιβαία να ε, μειώνονται όλο και περισσότερο οι μισθοί ε, ε, χωρίς κρατική υποστήριξη δεν μπορεί να επιβιώσουν τα αεροδρόμια. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε με μηδενικά τέλη να λειτουργήσουμε. Τώρα, εις ό,τι αφορά τους ε, κατοίκους, ε, ιδιαίτερα οι παρακείμενοι υποφέρουν όλο και περισσότερο από την αυξημένη κίνηση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και τις επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο. Το άρθρο 10 για την αρμοδιότητα ελέγχου της Κομισιόν πρέπει να απορριφθεί ο περιορισμός ε, της λειτουργίας θα πρέπει να είναι το πρώτο μέτρο ούτως ώστε η θυγόμενη περιοχή να θωρακιστεί και να προστατευτεί από τον θόρυβο. Η υγεία προέχει του οικονομικού του κέρδους. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα Θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Περόνη της Ομάδας για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με ε, τα σλότ, της χρονοθυρίδες, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν ένα μέσο διατήρησης των πλεονεκτημάτων και κάποιων κεκτημένων θέσεων αλλά θα πρέπει να είναι μέσο το οποίο θα ευνοήσει τον ανταγωνισμό διευκολύνοντας και άλλες αεροπορικές επιχειρήσεις και κυρίως διευκολύνοντας τους επιβάτες. Ένα άλλο θέμα θα έλεγα είναι ο θόρυβος. Είναι αλήθεια ότι όσοι ζουν, όσοι κατοικούν κοντά σε αερολιμένες δεν θα πρέπει να υποφέρουν από το θόρυβο. Θα πρέπει όμως θα έλεγα να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η συγκυρία. Θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο ε, του περιβάλλοντος χώρου πόσοι κατοικούν γύρω από το, το αεροδρόμιο οι οποίοι γνώριζαν ίσως οι περισσότεροι ε, τι σημαίνει η λειτουργία ενός αεροδρομίου. Η κυρία Φώστερ Σήκωσε την μπλε κάρτα της. Δέχεστε. Έχετε το λόγο κύριε Φώστα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σπερώνη αν συμφωνεί μαζί του όταν συζητάμε το θέμα του θορύβου ότι κάποιοι χαλαροί πολιοδομικοί κανόνες από πλευράς κυβερνήσεων και τοπικών αρχών αυτά τα χρόνια είναι μία από τις βασικές αιτίες για τον θόρυβο ο οποίος επηρεάζει τις περιοχές κατοικίας που είναι κοντά σε αερολιμένες. Νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να μην μπορούν να δίνουν άδειε για οικοδόμηση τέτοιων κατοικιών όπου το επιθυμούν χωρίς έλεγχο στο μέλλον. Ναι, κοιτάξτε, αναφερθήκατε στις τοπικές αρχές. Πράγματι σε κάθε χώρα ε, λειτουργεί διαφορετικά, γιατί σε κάθε χώρα είναι διαφορετική η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδεια ε, σε επίπεδο πολεοδομικό. Θα ήθελα όμως να κάνω εδώ μια σκέψη αν θέλετε. Ε, εντάξει, πράγματι μπορεί να εκδώσει μια άδεια μια τοπική αρχή. Παρ' όλα αυτά ενδιαφέρεται η τοπική αρχή για το αν θα κτίσει και αν θα πάει να κατοικήσει κάποιος κοντά στο αεροδρόμιο. Οι τοπικές αρχές δεν υποχρεώνουν κάποιον να πάει να κατοικήσει κοντά στο αεροδρόμιο. Ευχαριστώ. Είστε επαγγελματία στον χώρο αυτό κύριε Σπερώνη και ξέρετε γιατί μιλάτε. Λοιπόν, από πλευρά των μη εγγεγραμμένων έχει το λόγο ο κύριος Μέλτσερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι εποχές για τα αεροδρόμια, προστίθενται αεροπορικές εταιρείες, αυξάνεται το κόστος κυροζήνης, ε, όλοι ε, έχουν ελλείμματα παρά, τις, ε, παρά ε, την, την αύξηση ε, των επιβατών. Τα μικρά αεροδρόμια περιορίζουν την κίνηση και πολλές φορές οι συνθήκες είναι απαγορευτικές. Ένα άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών, οι εδάφους, θα οδηγήσει όμως σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το αμφιβάλλω. Οι μέχρι τούδε εμπειρίες δείχνουν ότι οι προσπάθειες απελευθέρωσης δεν έχουν πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμα και αν οι ρυθμίσεις δεν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα αεροδρόμια. Και σίγουρα πρέπει να εμποδίσουμε το μισθολογικό dumping. Μια καλύτερη αξιοποίηση των σλότς ε, ε, ε, επί απογείωσης και προσγείωσης είναι σημαντικό. Όμως με την προτινόμενη ρύθμιση για τις χρονοθυρίδες αμφιβάλλω αν θα επιτύχουμε το αποτέλεσμα αυτό. μπλε κάρτα από τον κύριο Λάιτφριντ. Αλλά δεν είναι η σύγγινης ο κύριος Λάιτφριντ. Όχι κύριε Λάιτφριντ. Σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κάρτα για τους συναδέλφους οι οποίοι περιλαμβάνονται στη συζήτηση μέχρι τώρα κλείσαμε με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων και περνάμε τώρα στους ομιλητές. Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Όλο το πακέτο για τα αεροδρόμια νομίζω ότι έχει αποτύχει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό σε καθοριστικά σημεία έχει βγάλει κάποια δηλητηριώδη δόντια, καμιά φορά και όλη την οδοντοστοιχεία. Ε, υπάρχει το θεμητό πρόβλημα ε, των πολιτών ότι η Κομισιόν ανακατεύεται πολύ περισσότερο από όσο πρέπει. Εμείς μειώσαμε το ρόλο της Κομισιόν. Ναι, ε, θα ενημερώνεται για τους περιορισμούς, ε, αλλαγές, θα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της, αλλά όχι ε, υποχρεωτικά και αυτό είναι σημαντικό. εκεί όπου δημιουργείται ο θόρυβος, εκεί πρέπει και να αντιμετωπίζεται. Ε, ε, θα πρέπει επιτέλους να αποσυρθεί η πρόταση όπως είπε η Επιτροπή Μεταφορών. Δεν επιτυγχάνει μεγαλύτερη ποιότητα η ύπαρξη περισσότερων παρόχων γιατί δημιουργούνται περισσότερες διαδικασίες εν κενό και μειώνεται η παραγωγικότητα εργαζόμενο. Εσείς δεν μας αποδείξατε ότι ένα απελευθερωμένο αεροδρόμιο λειτουργεί καλύτερα από ότι ένα αεροδρόμιο με δύο παρέχοντας μόνο. Το απελευθερωμένο κομμάτι των υπηρεσιών εδάφους δείχνει για τους υπόλοιπους πού πηγαίνει η κατεύθυνση εις ό,τι αφορά τους μισθούς. Ε, και αυτό δεν το θέλουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνωμοδότηση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Επιτροπής Μεταφορών σε αυτό το θέμα, αν μετά από μια απόρριψη και νομοθετικό ψήφισμα αρνητικό ε, μπορούμε να ξαναδούμε το φάκελο αυτό. Ε, μπορούμε να ε, εξετάσουμε δηλαδή μία πρόταση η οποία θα είναι πιο συγκεκριμένη και θα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας αφού αποσυρθεί η παρούσα πρόταση. Όχι όμως να απειληθούν οι μισθοί και να κάνουμε αναγκαστική απελευθέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φλέκενστάιν, δυόμιση λεπτά για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ένα διαδικαστικό. Μπορείτε να μου πείτε ε, ε, ποιο είναι το άρθρο του ιστορικού κανονισμού στο οποίο, το οποίο επικαλείστε για να ε, ζητήσετε διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να καταγράψω το εξής. Ε, προηγουμένως δέκα φορές ε, παρουσίασε μπλε κάρτα ένας συνάδελφος. Δεν πειράζει, όμως ε, πολλές φορές παρεμβαίνουν και μετά δεν περιμένουν την απάντηση και δεν έρχονται ήθελα ο κύριος Μέλτσερ εφόσον είναι ακόμη παρόν να μου απαντήσει κάτι αλλά δεν είναι εδώ και δεν πρόλαβα να του κάνω την ερώτηση διότι πολλοί ομιλούν και φεύγουν. Ε, συγγνώμη, αναγνωρίζετε κι εσείς ότι δεν είναι διαδικαστικό το ζήτημα που θέσατε. Σας σέβομαι και σας άκουσα μέχρι τέλους. Όμως ε, ε, τα άρθρα του εσωτερικού κανονισμού προβλέπουν ε, τη διαδικασία για τα διαδικαστικά και δεν πληρούνται τώρα τα κριτήρια. Έχουμε τη διαδικασία της μπλε κάρτας και είναι παρεμφερής της διαδικασίας Catch the Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών και δεν μπορούμε παρά να είμαστε αυστηροί διότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος αγόρευσης για όλες τις πολιτικές ομάδες και δεν μπορούμε να δίνουμε το λόγο σε όλους όσους δεν αναγνωρίζουν καταγράψει στον κατάλογο. Θα ακούσουμε τον κύριο Κνούτ δύο μισή λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και καιρό μιλάμε για τις υπηρεσίες εδάφους και ο κύριος Ζασάντα έχει δίκιο. Η απελευθέρωση άρχισε πράγματι το 1996, αλλά είχε μοιραίες συνέπειες για τις αμοιβέ και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Στο επίκεντρο του σημερινού κανονισμού βρίσκεται ένα μέτρο το οποίο ε, υποχρεώνει και έναν τρίτο ανταγωνιστή. Ε, ε, ε, τυπικά γιατί επί της ουσίας υπάρχει και ρίξαμε λάδι στη φωτιά προσθέτοντας και έναν τέταρτο δεν θα το δεχτούμε αυτό οι σοσιαλδημοκράτες λένε ότι χωρίς αντίστοιχη διασφάλιση των εργαζομένων δεν γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή ρυθμισμένη μεταβατική περίοδος για όλους ε, αντιπροσωπευτική συλλογική σύμβαση ελάχιστοποίηση του αριθμού των υπεργολάβων ε, και η όροι του παιχνιδιού. Αυτά δεν εξασφαλίζονται και γι' αυτό δεν μπορεί να δεχτούμε περαιτέρω αναγκαστική απελευθέρωση. Επίσης δεν είναι εφεύρημα γερμανοαυστριακό αυτό, αλλά είναι το συμπέρασμα του Συνδικάτου των Εργαζομένων στις Μεταφορές. Ο στόχος της αυξημένης ανταγωνιστικότητα, των, ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, ε, κατά τη γνώμη μου, δεν επιτυγχάνεται με το μέτρο που προτείνεται. Και επιτρέψτε μου να πω ένα πράγμα, κύριε Επίτροπε, στη European Voice αναφέρεστε, υπάρχει ένα παράθεμα, ότι είστε ε, απογοητευμένος γιατί οι αεροπορικές εταιρείες δεν έκαναν αρκετό ενεργό ακτή ε, lobbying ε, και το αναφέρει και στα αγγλικά το παράθεμα στα αγγλικά ε, σπάνια συμβαίνει συνάδελφοι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βλέπει ένα σχέδιο να του επιστρέφεται γιατί δεν είναι καλό και μετά να λυπάται διότι οι ευνοημένες ε, επιχειρήσεις δεν άσκησαν επαρκή επιρροή. Και πρέπει να σας πω κύριε Επίτροπε ότι αυτό είναι λάθος γιατί όλες ήρθαν να με βρουν αλλά δεν με πείσανε. Ε, οι λόμπις ε, που με ε, ενημέρωσαν είναι οι Μούλερ, Κόβατς, Τζοντζάλε, Σμιθ και με πάνω από 3.000 συναδέλφους ήρθαν εδώ έξω από το κοινοβούλιο γιατί φοβούνται για τις άσχημες συνθήκες εργασίας τους. Αυτοί μάλιστα με έπεισαν ότι δεν επιτρέπεται να δεχτούμε την πρόταση που μας υποβάλλεται. Ευχαριστώ. μία ερώτηση στα πλαίσια της μπλε κάρτας, ο κύριος Ζασάντα. Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να τη και δίνω το λόγο στον κύριο Πίρκελ. Θέλετε να απαντήσετε στον συνάδελφο Πίρκελ. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Κύριε Φλέκενστάιν, ε, επί της ουσίας ε, συμφωνώ με τις απόψεις σας εις ό,τι αφορά τις υπηρεσίες εδάφου. Το ερώτημα είναι όμως ποιες είναι οι λογικές συνέπειες από το συλλογισμό σας ε, και ερωτώ εσάς και την ομάδα σας αύριο την, πρόταση, την νομοθετική πρόταση θα την απορρίψετε στη, κατά τη συνολική ψηφοφορία όπως είχε προτείνει η Επιτροπή η αρμόδια επιτροπή. Μάλιστα. Ε, σαφής η ερώτηση, σαφής και η απάντηση. Ναι, αυτό προτίθεμε να κάνω. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Τρεμός θα έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ε, καλή δουλειά και ευχαριστώ και τον φίλο Γιώργ Λάιχτφριντ. Θα τα πω αγγλικά. Δεν είναι καλά τα γερμανικά μου. Ε, το άρθρο για το δικαίωμα εξέτασης ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα θετικό στοιχείο και υπάρχει παρανόηση νομίζω. Ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα ε, κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα για τους Γερμανούς συναδέλφους ε, που είναι παρόντες σήμερα. είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τη διαδικασία και ουχή το περιεχόμενο, ούτε καν τις τοπικές αποφάσεις. Δίχως αυτό το μέτρο εκτίθενται οι φορείς ε, στο ενδεχόμενο αυθαίρετης και διακριτικής διαδικασίας επιλογής για την κατανομή χρονοθυρίδων βάση των πινάκων που κατέθεσαν το ΕΛΚ ε, και, το, εκεί οι σοσιαλιστές 44 ε, και 48 για τα άρθρα 1 και 2 ε, θα δώσω τη σύμφωνη γνώμη μου διότι σε αυτές τις τροπολογίες αναφέρουμε το θέμα του κόστους και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ανέκαθεν το υποστήριζαν αυτό οι φιλελεύθεροι και με αυτήν την τροπολογία βελτιώνεται το κείμενο. Όμως σημειώστε ότι οι τροπολογίες 45 και 49 Πλημελώ ε, κατά τη γνώμη μου αυτή την εξορροπημένη προσέγγιση. Ο μετριασμό ε, του θορύβου σημαίνει ότι η χωμόνωση στα σπίτια ε, καθώς και τα μέτρα αλλαγή χρήση γη, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν γιατί δεν είναι άμεσα μέτρα μετριασμού θορύβου. Σα ευχαριστούμε κύριε Τρεμόσα. Ε, ε, Μίχαλ Κράμερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Κάλλας, χάρηκα που συμπεριλάβατε το θέμα του θορύβου. Αλλά όπως στις εκπομπές νομίσαμε ότι θα υπάρξουν ελάχιστα όρια που δεν μπορεί κανείς να υπερβαίνει. Ε, δεν έγινε όμως αυτό το πράγμα. Εσείς ως Κομισιόν ε, θέλετε να αποφασίζετε για το θόρυβο και τις συνέπειες που αυτός ε, δημιουργεί. Φανταστείτε μια πρωτοβουλία πολιτών στη Γερμανία που δίνει μάχη για τη μείωση του ε, θορύβου που πείθει την τοπική βουλή, την κρατηδιακή βουλή ε, και προβαίνει σε, νυχτερινές, σε απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων. Και εσείς ε, πάτε μετά ως Κομισιόν και λέτε όχι θα το αλλάξουμε αυτό, εμείς ε, θα αποφασίζουμε, έρετε η απαγόρευση των πτήσεων. Δηλαδή χειρότερο δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι αντιευρωπαϊκή θέση. Είναι πολύ άσχημο και καλό είναι που ε, αποσύρθηκε η πρόταση. Θέλουμε όμως γνωμοδότηση και ε, ε, ενδεχομένως τα δικαστήρια μπορεί να αποφανθούν ότι ε, έχει δίκιο η Κομισιόν, δηλαδή ότι το κέρδος μας ενδιαφέρει και όχι ο κόσμος. Αν πρόκειται για τα λεφτά, σας το ξαναλέω, οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη κάθε χρόνο από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους παίρνουν 30 δις ευρώ δώρο γιατί ε, δεν πληρώνουν φόρο κυροζήνης και προστιθέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει ότι τα πληρώνουν όλα οι ε, καταναλωτές. Ε, φανταστείτε, ε, αν αυτά τα έπαιρναν οι, τράπεζες θα είχαμε ε, καλύτερο δίκτυο και καλύτερες υπηρεσίες και δεν θα είχαμε αυτό τον κορεσμό στις εναέριες μεταφορές όπως είπατε εσείς. Είναι φούσκα αυτή όπως τα ακίνητα στην Ισπανία. Δεν μπορούμε να την ανεχθούμε και στις εναέριες μεταφορές. Θέλουμε θεμητό ανταγωνισμό, ε, σωστές δίκαιες τιμές. Δεν μπορεί οι μένα πληρώνουν και οι άλλοι όχι. Και δεν μπορεί αυτοί που καταστρέφουν το κλίμα να ε, ε, επενούνται και να καταστρέφονται οι άλλοι. Γιατί αυτό είναι που προδιαγράφεται για την Ευρώπη. πάση περιπτώσει δεν έχω παρακολουθήσει το τι έλεγε ο μετρητής του χρόνου ε, και γι' αυτό είχατε δυνατότητα να εκφραστείτε, αλλά ελπίζω χωρίς ε, να περιοριζόμαστε κάπως χρονικά στο μέλλον. Παντάλεν, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να ωφεληθεί από την ενιαία αγορά, από την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των προσώπων. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι ισχύ και οι οποίες βασίζονται, δράζονται σε ιδέες μονοπωλίου και σε ιδέες προστατευτισμού. Αυτό ισχύει για τον τομέα σαν παράδειγμα της, ε, της ε, εξυπηρέτησης εδάφους των υπηρεσιών εδάφους. Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Το θέμα είναι βέβαια να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε την αγορά από ό,τι φαίνεται τα συνδικάτα έπεισαν κάποια μέλη και η πρόταση αυτή θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Θα έχουμε χάσει μια ευκαιρία. Γιατί θα έχουμε κάποια επιπλέον εμπόδια τα οποία θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις, τις αεροπορικές εταιρείες και θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις κυρίως για τους χρήστες των αεροδρομίων, τους ε, καταναλωτές η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να προτείνει ακόμα περισσότερα μέτρα για το άνοιγμα αυτών των αγορών. Ελπίζω αύριο να αντιμετωπίσουμε στην Ολομέλεια την πρόταση αυτή με σωστό τρόπο. Μια πρόταση η οποία θα μας δώσει την δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε και θα πρέπει να επανέλθουμε με τον τρόπο που πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Δύο έχουν ζητήσει την μπλε κάρτα. Το ένα ο κύριος Γκάλερ που δεν του δώσω το λόγο γιατί έχει ήδη σηκώσει, έχει ήδη μιλήσει και το άλλο για τον κύριο Λιμπεράτσκι. Κοιτάξτε, αν θέσετε ερώτημα δεν θα μιλήσετε μετά. Τι προ... Με μικρόφωνο δεν σας ακούμε. Ε, διαλέγω να μιλήσω για 90 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Κύριο Σκόχλιτσεκ. Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος εναερίου ελέγχου, υπάρχει ανάγκη αύξησης της χωρητικότητας ορισμένων αερολιμένων και να τροποποιήσουμε δηλαδή τους όρους λειτουργίας των αερομεταφορών, ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες ε, εποχές του χρόνου. Αυτό θα ελαφρύνει γενικά ε, κάποιες καταστάσεις ε, κορεσμού οι οποίες παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή λειτουργία ενός Ευρωπαίου συντονιστή και θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ανεξαρτησία των εθνικών συντονιστών. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή θα ήταν η καλύτερη και ένα σχόλιο να κάνω για τον κύριο Βαντάλεν. Νομίζω ότι τα συνδικάτα ε, είναι ψηφοφόροι σας. Μην το ξεχνάτε αυτό παρακαλώ όταν συζητάτε τέτοια θέματα γιατί μπορεί να μην επανεκλεγείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πακέτο για τα τσαρολιμένες, οδήγησε σε πολλές συζητήσεις και ως συντονιστής του ΕΛΚ δεν είχα εύκολη δουλειά να κάνω. Τα ακούσατε, γι' αυτό θα ήθελα ε, να δούμε με κάποιες αποχρώσεις ε, το θέμα αυτό. Ε, σε ό,τι αφορά το θόρυβο, γενικά νομίζω ότι το έργο ήταν καλό. Ευχαριστώ όλους τους συζητητές γιατί... Ε, λαμβάνουμε υπόψη με δίκαιο τρόπο τα πράγματα και σεβόμεθα πολλές ε, συμφωνίες ε, που έχουν γίνει εις ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και με τους κατοίκους. Εγώ προέρχομαι από μια ε, περιφέρεια όπου όλα αυτά στήχησαν εκατομμύρια και όλοι ε, μπόρεσαν να καλυφθούν από μια πολύ καλή συμφωνία. Αυτό είναι ο στόχο, να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Σε ό,τι αφορά τα χρονικά περιθώρια, θα ήθελα μια βελτίωση, γιατί το σημαντικότερο για μένα, α, το, με τι χρονοθυρίδε, συγγνώμη, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, γίνει βέλτιστη χρήση του και να υπάρχει και διαφάνεια. Ε, τώρα για τις υπηρεσίες εδαφούς θέλω να πω το εξής. Αν δείτε τι είχαμε συμφωνήσει το 1996, ε, τότε δεν υπήρχαν ελάχιστα πρότυπα ποιότητας ούτε πρότυπα για την εκπαίδευση κατάρτιση, ούτε για την ε, μετεκπαίδευση επιμόρφωση. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία, και αυτό πρέπει να πούμε στους 3.000 ε, που είναι έξω, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία, τότε και το λέει ε, η καταπλειοψηφία το ΕΛΚ πρέπει να πάει ο φάκελο στην Επιτροπή πίσω για να τύχει επεξεργασία και βελτιώσεων. Αυτή είναι η ευκαιρία μας. Και δεν πρόκειται για δραστική αύξηση της αγοράς, μεγέθυνση της αγοράς, όταν έχουμε απελευθέρωση από τους δύο στους τρεις που αυτό αφορά ε, ελάχιστα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό ε, ε, είναι σημαντικό να το πούμε και να είναι και σωστή η ενημέρωση. Αυτή τη συζήτηση ήθελα να την κάνουμε και όταν μιλήσαμε όταν μιλούσαμε και για την οδηγία για τις ταχυδροπικές υπηρεσίες. Εκεί δεν είχαμε μεγάλη ευαισθησία για τις εργασιακές συνθήκες. Εδώ ε, είναι πιο, οξυμένο, πιο οξυμένη η συζήτηση. Πιστεύω λοιπόν ότι μια καλή συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα και θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους. Έκλεισε το μικρόφωνο του ομιλητή. Κοιτάξτε, δεν έχετε άλλο χρόνο πλέον. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο σας. Για δυόμιση λεπτά ο κ. Σασόλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μια πολύ σημαντική δραστηριότητα μεταφορική. Αύριο τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και τα πράγματα σίγουρα θα γίνουν πιο δύσκολα γιατί οι κανόνες μας, οι υποδομές μας ε, δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ε, ζήτηση. Το κείμενο το οποίο θα κληθούμε να ψηφίσουμε αύριο περιλαμβάνει ορισμένες μικρές βελτιώσεις, επιμέρους βελτιώσεις και κάποιους τοπικούς κανόνες που θα επιτρέψουν στα αεροδρόμια να έχουν μεγα, μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο κατανομής και χρήσης των χρονοθυρίδων. Μια καλύτερη εκμετάλλευση της αγοράς των αερολιμενικών εγκαταστάσεων ε, και μέσω της δευτερογενούς αγοράς των χρονοθυρίδων από την άλλη βέβαια το κείμενο ως έχει μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη ψυχραιμία θα έλεγα και γαλήνη. Αλλά εγώ θα ήθελα εδώ να πω ότι απαιτείται μεγαλύτερο θάρρος, περισσότερο θάρρος, θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξουν πιο σημαντικές αλλαγές, πιο ουσιαστικές αλλαγές θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της σωστής ε, ε, χρήσης ε, των δυνατοτήτων που έχουμε στον τομέα τον αερολιμενικό σύμφωνα με τον κανόνα που λέει ότι αν δεν το χρησιμοποιείς θα το χάσεις σχετικά με τις χρονοθυρίδες. Use it or lose it στα αγγλικά. Και η αναθεώρηση των κανόνων θα πρέπει να γίνεται κάθε 8 ή 10 χρόνια γιατί μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν πολύ γρήγορα στις αερομεταφορές. Απαιτείται θάρρος λοιπόν περισσότερο και γι' αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο σημαντικά βήματα επιβάλλοντας πιο ορθολογικούς κανόνες, πιο μακροπρόθεσμους κανόνες και με καλύτερα θεμέλια από αυτά τα οποία προτείνουμε σήμερα. Κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Το αποτέλεσμα καλό είναι, αλλά δεν είναι το καλύτερο δυνατόν. Σίγουρα το κείμενο δεν είναι κακό, η πρόταση δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι και ό,τι περιμέναμε. Κυρία Μάσινα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν συναισθηματικά φορτισμένη η συζήτηση. Σπάνια το διάστημα που είμαι στο Κοινοβούλιο. Ε, επιδιώκουμε περισσότερα. Όλη η πρόταση για το πακέτο των αερολιμένων ε, σκοπό είχε να ε, προετοιμάσει το Single European Sky, ενιαία η Ευρωπαϊκή Ουρανή και να βελτιώσει την κατάσταση για το θόρυβο είπαμε ότι δεν πρέπει να ε, παίζουμε την υγεία σε αντιπαράθεση με το κέρδος. Αν δούμε μόνο την υγεία όμως και δεν δούμε πώς λειτουργούν τα ιερολιμένες, αυτό δεν είναι εξισορροπημένη προσέγγιση που όμως τι θέλουμε. Γιατί θέλουμε η οικονομία να ανθεί και στους αερολιμένες και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες εδάφους. Πραγματικά, όπως ο Ματιό Εγκρός, η απελευθέρωση ήταν παλιότερα δυνατή. Μεγάλα αεροδρόμια με δύο παρόχους είχε καλή ποιότητα. Αυτό δεν ισχύει παντού. Αλλά δεν ε, είχαμε πρότυπα εξειδίκευσης για την απασχόληση και την κατάρτιση των εργαζομένων. Αυτό είναι κάτι που τώρα όμως μπορούμε να το ξαναδούμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ζαμπέλ Τυρό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το να θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών στα αεροδρόμια είναι θεμητό, αλλά τώρα οι επιπτώσει συγχωρήπανση επί της υγείας δεν χρειάζεται να καταδειχθεί. Δεν είναι θέμα άνεση όπω προσπαθούν να μα πείσουν κάποιοι. Είναι ένα θέμα υγεία και πρόορου θανάτου σε ορισμένες περιπτώσεις. Κυρία Μάισνερ, θέλουμε μια σωσκελισμένη πρόταση. Υπάρχουν και οι προτάσει του... Ε, δεν ενσωματώνουν οι προτάσει του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία, άρα δεν είναι εξισορροπημένη η πρόταση λυπάμαι πολύ. Ε, αυτό που ζητάμε είναι να ισχύει ένα ενιαίο κανόνα, ούτω ώστε η Επιτροπή να μην έχει τη δυνατότητα ε, να αναιρέσει αυτά που οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ με δυσκολία ε, έχουν καταφέρει. Δεν καταλαβαίνω τι σα ενοχλεί το να περάσουμε από δύο σε τρει παρόχου. Αν η απελευθέρωση μα βοηθάει να καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικέ υπηρεσίε, πρέπει να το καταδείξουμε στον τομέα των μεταφορών και δεν καταλαβαίνω με ποιο τρόπο ενισχύουμε την αύξηση του αριθμού των παρόχων την ποιότητα των υπηρεσιών. Ε, εάν ε, θα πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση μόνο να αναπευθεί στην αρμόδια επιτροπή. Ευχαριστούμε, Ιζαμπέλ. Ο κύριο Τούσα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που συγκροτήθηκαν και κυριαρχούν στι αερομεταφορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατούν σε αυξήσει φωτιά στι τιμέ των εισιτηρίων επιβατών και εμπορευμάτων, στη μείωση τη συχνότητα των αεροπορικών δρομολογίων, μαζικέ απολύσει, εντατικοποίηση τη δουλειά και δραστικέ μειώσει στους μισθού των πληρωμάτων των αεροπλάνων και των εργαζομένων στις υπηρεσίες εδάφους διαλύουν τι εργασιακέ σχέσει, υποβαθμίζοντα συνολικά τι αεροπορικέ υπηρεσίε. στην ελλάδα ο επιχειρηματικό όμιλο που μονοπολεί την αγορά μετά το ξεπούλημα τη Ολυμπιακή κατάργησε το τμήμα υπηρεσιών εδάφου και μετέφερε όλο το προσωπικό της 850 άτομα στην gold air handling τη μεγαλύτερη σήμερα εταιρεία του κλάδου προχωρώντας σε μειώσεις μισθών μαζικές απολύσεις και εντατικοποίηση της δουλειάς. οι εργαζόμενοι αντιπαλεύουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που αποσαφρώνει εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις κάνει πανάκριβες για το λαό της αερομεταφορές χειροτερεύει την ποιότητα των υπηρεσιών και βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών. στην αντιλαϊκή πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεων οι εργαζόμενοι προτάσουν τη δική τους λύση για σύγχρονες φτηνές αεροπορικές μεταφορές για το λαό με πλήρη δικαιώματα για τους εργαζόμενους του κλάδου και προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. λεπτά. Κυρίες και κύριοι, η πρόταση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει προωθήσει την ποιότητα, προσπαθεί να διευκολύνει τον επιβάτη. Θα πρέπει να βελτιωθεί η παροχή των υπηρεσιών, είναι βασικός στόχος. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χωρατικότητα των αεροδρομίων Θα πρέπει επίσης να διαχειριστούμε καλύτερα και το θέμα του θορύβου από πλευράς των αεροπλάνων στις περιοχές γύρω από τα αεροδρόμια που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Και θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και τις ε, υπηρεσίες ε, που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία και εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία τίθενται και ο συνάδελφος ο Ζασάντα έχει δίκιο όταν ζητά να υπάρξει περισσότερος χρόνος έτσι ώστε η Επιτροπή Μεταφορών να βρει μια λύση η οποία να είναι ικανοποιητική για όλους. Σίγουρα υπάρχουν συμφέροντα νόμιμα τα οποία ε, εκφράζονται γύρω από το θέμα αυτό αλλά απαιτείται χρόνος, απαιτείται συνοχή πολιτική και φυσικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι κατά της απελευθέρωσης, είναι κάτι το οποίο όμως δεν θα πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων. Νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε με ευθύνη και δεν θα πρέπει να υπακούσουμε σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι όλα θα αλλάξουν όταν δεν αλλάξει τίποτα. Για δύο λεπτά το λόγο έχει πλέον η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα πλαίσια της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων εξετάσαμε την πρόταση αυτή με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το οποίο μας κάνει πραγματικά εντύπωση είναι ότι τη στιγμή που σοβεί η συγκεκριμένη κρίση, τη στιγμή που η πλήρης φιλελευθεροποίησης έχει καταστρέψει τεράστια κομμάτια της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται με μια πρόταση φιλελευθεροποίησης για μια ακόμη φορά λέγοντας ότι οι υπηρεσίες που θα δίδονται στους επιβάτες θα έχουν καλύτερη ποιότητα και μειωμένη τιμή. Κοιτάξτε, βλέποντας τις υπηρεσίες στους αερολιμένες δεν είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της πρότασης τη Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει και έχουμε καταθέσει εκ νέου ορισμένε τροπολογίε στην περίπτωση κατά την οποία η πρόταση απόρριψη τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέθεσε ο κ. Σίμψον δεν ψηφιστεί από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Θα καταθέσουμε εκ νέου λοιπόν τις τροπολογίες που είχαμε κάνει δεκτές στην αρμόδια επιτροπή για να εμείνουμε σε ορισμένα σημεία τα οποία θεωρούμε βασικά. Το ένα είναι το θέμα της μεταφοράς των δικαιωμάτων των εργαζομένων όταν υπάρχει μεταφορά από επιχείρηση σε επιχείρηση, απώλεια άδεια εκμετάλλευση ή τροποποίηση παροχής υπηρεσιών. Όταν ο υπεργολάβος στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλάζει, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση να συνεχίσουν να χαίρουν των ιδίων εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό είναι αναπόσπαστο τμήμα θα έλεγα Τη λογική που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει το θέμα τη ασφάλεια, τη υγεία, στον χώρο απασχόληση, τη καταπολέμησης του μισθολογικού ντάμπινγκ. Φοβόμαστε ότι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι όπω προτείνεται από την Επιτροπή θα μα οδηγήσει σε μια χειροτέρευση τη κατάσταση του επίπεδου εργασία του προσωπικού ε, των αεροδρομίων που θέλετε για μια ακόμη φορά να φιλελευθερωποιήσετε. Ευχαριστώ Περβάνς. Η κυρία Σαβισάρ το Μάστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Ε, φυσικά πρέπει να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότερα μεταφορά επιβατών και φορτίου. Ταυτόχρονα όμως ε, με τους νέους κανονισμούς ε, δεν πρέπει να βρεθούν σε χειρότερη θέση κάποιες επιχειρήσεις, κυρίως οι μικροί φορείς διαχείρισης αεροδρομίων. Οι τροπολογίες 26 και 83 στην έκθεση για τις χρονοθυρίδες με απασχόλησαν ιδιαίτερα. Η πρώτη υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία. Και η 83 ουσιαστικά νερή την 16. Εγώ συμφωνώ ότι είναι προβληματική η κατάσταση με τις χρονοθυρίδες και δεν ε, χρησιμοποιούνται ε, αποτελεσματικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των ε, ενδιαφερομένων. όταν ένας φορέας ε, ε, μπορεί να χρησιμοποιεί τις χρονοθυρίδες αλλά όχι συναπτά δεν χάνει το δικαίωμα που έχει στους χρονοθυρίδες και πιστεύω ότι αυτό δεν συνιστά αποτελεσματική χρήση των ε, σλότς. Ε, θα έπρεπε λοιπόν ε, στην οδηγία για τις χρονοθυρίδες να υπάρχει μια τακτικότητα στα μέτρα που προτείνουμε. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτό κύριο Σπίρκερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το θέμα είναι τι περιμένουν οι επιβάτες από τις υπηρεσίες εδάφους να, έρθει, να έρθουν οι αποσκευές, να πιούν κάτι, να είναι ασφαλείς, γιατί δεν τους πειράζει, δεν ενδιαφέρονται για το πώς αισθάνει οι υπηρεσίες, οι εταιρείε υπηρεσίας εδάφους η ρύθμιση που υπάρχει επιτρέπει ευέλικτη διαχείριση. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο. Η απελευθέρωση είναι δυνατή. Μπορεί να είναι τρει, μπορεί να είναι πέντε, μπορεί να είναι και δέκα. Και οι αερολιμένες στην Ευρώπη αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Γιατί κάποια, ε, κάποιοι αερολιμένες έχουν δύο, άλλοι περισσότεροι. Περισσότεροι πάροχοι δεν σημαίνει ταυτόχρονα ε, ότι υπάρχει εγγύηση λειτουργίας των υπηρεσιών. Έχουμε παραδείγματα όπως στη Βιέννη για παράδειγμα όπου ε, δύο εταιρείε εγγυώνται ακρίβεια και ποιότητα 99%. Υπάρχουν άλλοι αερολιμένες με τέσσερις εταιρείε και δεν είναι ικανοποιημένοι οι επιβάτες με τις υπηρεσίες που παρέχονται. Δηλαδή οι περισσότερες υπηρεσίες δεν σημαίνει αναγκαστικά και καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή τώρα τι, ποια είναι η θέση μου. Η ρύθμιση σήμερα επιτρέπει την απελευθέρωση. Δεν βλέπω προστιθέμενη αξία με την υποχρεωτική περαιτέρω απελευθέρωση. Δηλαδή να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε τρεις, οπωσδήποτε τέσσερις εταιρείε με τις δύο κατελάχιστον. Έχουμε ανταποκριθεί στο στόχο της απελευθέρωσης και βλέπουμε ότι είναι μια πολύ λειτουργική ρύθμιση αυτή για τους αερολιμένες. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στο Κοινοβούλιο αύριο να ακολουθηθεί η πρόταση της Επιτροπής για την αναπομπή της πρότασης της Κομισιόν και παρακαλώ τον κύριο Επίτροπο μετά από την ψηφοφορία αυτή να αποσύρει και εκείνο την πρότασή του. Δύο λεπτά και για την κυρία Στάινροκ. Και εμείς οι σοσιαλδημοκράτες ενδιαφερόμεθα για την οικονομική ευρωστία της Ευρώπης. Αλλά για να υπάρχει αυτό πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι, με καλά κίνητρα οι εργαζόμενοι, ε, καλά καταρτισμένοι. Πήραμε πληροφορίες από τα συνδικάτα σχετικά με τις επιπτώσεις της περαιτέρω απελευθέρωσης της υπηρεσίες εδάφους. Ε, και γι' αυτό είμαι απογοητευμένη γιατί όταν έχουμε εδώ απ' έξω ε, μια εταιρεία ε, οικονομικού, οικονομικών συμφερόντων δεν έχω δει ε, ε, τέτοια, ε, δια, τέτοιες διαμαρτυρίες όπως ακούσαμε για τους εργαζόμενους ο, κύριε Επίτροπε, κύριε Σασάντα συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα η πολιτική απελευθέρωση τι ε, δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται για τη θέση εργασία του, φοβούνται ότι στο μέλλον δεν θα μπορούν να θρέφουν πια τι οικογένειε του, φοβούνται τι ανασφαλεί επισφαλεί θέσεις εργασίας. Είναι κρίμα αυτό που <clears throat> συμβαίνει. Να σκέφτεστε και την οικονομία βεβαίως, αλλά να σκέφτεστε και τα αποτελέσματα των προτάσεών σας και αν πάτε στον κόσμο και αν δείτε και τα νούμερα μάλιστα η κατάσταση μετά την τελευταία απελευθέρωση στη Γερμανία ε, οδήγησε σε μείωση 20% του πραγματικού μισθού 40% ε, ε στον τομέα των αερολιμένων. Ε, ε οι μισθοί πια δεν μπορούν να είναι αξιοπρεπείς και υπάρχουν και χώρες που η απελευθέρωση προχώρησε ακόμα περισσότερο και είναι ακόμα πιο ακραία τα αποτελέσματα. Βεβαίως χρειάζεται ανταγωνισμό, αλλά χρειάζεται και ποιότητα. Ποιότητα η οποία από ποιον εξασφαλίζεται, από τους ίδιους τους εργαζομένους αερολιμένες, τους οποίους δεν μπορούμε να τους ξεχνούμε στις προτάσεις μας. Ε, ε υπάρχει, ε, έγινε η προσπάθεια να ε, βελτιωθούν κάποια πράγματα, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν θέλουν ιστολογία οικοκοινωνικό κοινωνικό ντάμπινγκ, θέλουν καλή κατάρτιση, θέλουν προστασία. Ευχαριστώ. Κύριος σε 1,5 λεπτό. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία αυτής της ε, έκθεσης για τις υπηρεσίες εδάφους ε, στον τομέα των αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την σημασία των υπηρεσιών εδάφους εν γέννη, το να υπερψηφίσουμε την αναπομπή και ε, να ε, τοποθετηθώ υπέρ της αναπομπής της έκθεσης στην Επιτροπή. Χρειάζεται αυτή η έκθεση για να εξασφαλίσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό και την κατάλληλη ποιότητα για τις υπηρεσίες, τόσο για τους αερομεταφορείς όσο και για τους επιβάτες. Αυτό που μας απασχολεί εδώ δεν είναι μόνο η απελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφους. Μιλάμε επίσης για ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τους Ευρωπαίους πολίτες, για το τσέκιν και τη διακίνηση των αποσκευών τους. Επίσης δεν μιλάμε καθόλου εδώ για μέτρα που οδηγούν σε άγρια απελευθέρωση της αγοράς. Συζητούμε μόνο αύξηση του ελαχίστου αριθμού παρόχων από 2 σε ε, συζητούμε επίσης τα ελάχιστα πρότυπα κατάρτισης ε, για το προσωπικό του κλάδου καθώς ε, και για την προστασία των εργασιακών συνθήκων τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί εργάστηκε σκληρά. Ελπίζω όλοι σας αύριο να υπερψηφίσετε την αναπομπή στην Επιτροπή Μεταφορών αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 1,5 λεπτό έχει τώρα ο κύριος Λιμπεράτσκι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, γνωρίζω ότι έχετε καλές προθέσεις, αλλά καλές προθέσεις βρίσκει κανείς και στην κόλαση. Ε, θέλετε να αυξήσετε τη χωρητικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών ε, των αερολιμένων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους ε, παρόχους. Όμως δεν λαμβάνετε υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν σε κάποια τμήματα του κλάδου. Τι σημαίνει αυτό. Αν ακολουθήσουμε την δική σας πρόταση, εν τέλει θα είμαστε εντελώς αντιπαραγωγικοί. Ε, νομίζω Οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι εάν ένας εφορέας διαχείρισης έχει ένα μικρότερο ε, μερίδιο της αγοράς, πάσχει ο ανταγωνισμός και υπάρχουν ε, όλο ένα και μεγαλύτερα κενά. Δηλαδή, απασχολούμενοι εργάζονται λιγότερο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Άρα, ε, περιορίζεται η αποτελεσματικότητα ως προς το εργατικό δυναμικό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, θα περικόψετε τους μισθούς ή η αύξηση του αριθμού των παρόχων δεν ισούται με την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ορισμένες φορές δεν υπάρχει καν χωρητικότητα ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι τρεις και όχι οι δύο πάροχοι. Σας το Απέδειξε αυτό σήμερα και γι' αυτό ζητώ την αναπομπή στην Επιτροπή Μεταφορών και ε, απευθύνω έκκληση προς τους συναδέλφους, ε, κύριε Χίγκης, ε, κύριε Γκρός. Θα πρέπει να ψηφίσουμε για την αναπομπή της πρόταση, αλλά όχι στην Επιτροπή Μεταφορών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να προετοιμάσει ένα νέο σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τι ανάγκες όλων. Ευχαριστώ, Κόχ, επίσης για ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, ας αφήσουμε τους συναισθηματισμούς για να είμαστε ρεαλιστές. Ποτέ ένα ειδικό νομοθέτημα δεν ήταν σημαντικό όταν αφορούσε ελάχιστους εργαζομένους. Σήμερα μιλάμε για υπηρεσίες εδάφους που θα πρέπει υποχρεωτικά να απελευθερωθούν περισσότερο, αν και δύο πρέπει να είναι ο ελάχιστος αριθμός των εταιριών. Ε, πολλοί αερολιμένες δεν έχουν τρεις. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Ποιος αξιοποιεί αυτήν την ε, επίθεση στις δομές των αερολιμένων και αν οι ε, ευρωπαϊκές ε, αεροπορικές εταιρείες απειλούνται στην υπόστασή τους, τότε ανησυχούμε. Για να τις σώσουμε πρέπει να αρχίσουμε άλλες δραστηριότητες και μάλιστα άμεσα. Ε, διαγραφή της εμπορίας εκπομπών στις ενέργειες μεταφορές, ε, ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, ε, κατάργηση του φόρου καυσίμων στη Γερμανία. Υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότερα, αλλά γι' αυτό χρειάζονται πρότυπα, στάνταρ, καλύτερη επιμόρφωση, καλύτερη, καλή μισθή, όχι όμως αυθαίρετη αύξηση του αριθμού των παρόχων στην περιορισμένη αγορά. Παρακαλώ ψηφίστε αύριο υπέρ της πρότασης της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχετε πάρει ήδη το λόγο κύριε Κράμερ. Δίνω το λόγο για 1,5 λεπτό στην κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ό,τι αφορά τη μείωση του θορύβου και τις ε, χρονοθυρίδες, ε, ακούσαμε... Ε, ε, ενδιαφέρουσες προτάσεις για το θόρυβο. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ε, ε, θεμάτων οικονομικών και θεμάτων υγείας. Για τις υπηρεσίες εδάφους πρέπει να βελτιωθεί η χωρητικότητα και ο ανταγωνισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα για να γίνει ανταγωνιστική. Η απελευθέρωση όμως το, της αγοράς δεν πρέπει να είναι σε βάρος των κοινωνικών συνθήκων. Τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν τόσο το προσωπικό των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες εδάφους να προστατεύονται στον κοινωνικό τομέα και να έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Ε, και στα πλαίσια συμβάσεων παροχή υπηρεσιών. Και αν διαπιστωθούν κενά προστασίας ή αν παραδιάζονται πρότυπα, τότε η διαπίστευση αυτών των ε, παρόχων θα πρέπει να αναστέλλεται ή και να ε, διαγράφεται ή να ανακαλείται μέχρι να πληρούνται τα πρότυπα πάλι. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επαγρυπνούν για την τήρηση των ελάχιστων προτύπων για να δουν αν είναι αντίστοιχα εξειδικευμένο το προσωπικό και θα πρέπει να διασφαλίζονται μόνο υψηλά πρότυπα ασφαλεία, ελάχιστα πρότυπα για τις υπηρεσίε εδάφους θα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό το στηρίζουμε γιατί είναι καλό για τη λειτουργία των αεροδρομίων. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτοί οι οποίοι πήραν το λόγο πριν από μένα έθεσαν ορισμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ αποκλειστικά στο θέμα της επιβολής τιτικών ε, περιορισμών ε, για λόγους θορύβου. Στο τέλος του τελευταίου γύρου των συζητήσεων που είχε γίνει το 2002, από τότε έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει, ένα υπάρχει μια πολύ σημαντική επίπτωση στον τομέα της υγείας των κατοίκων γύρω από τις περιοχές των αεροδρομίων. Μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αυτοί οι οποίοι ζουν γύρω από τα αεροδρόμια φύγονται από τον θόρυβο, φύγονται σε επίπεδο υγείας, χάνουν την ακουστική τους οξύτητα τους δημιουργούνται και άλλα προβλήματα υγείας για λόγους τους οποίους οι ίδιοι δεν είναι υπεύθυνοι, δεν επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί να πάνε να ζήσουν στα αεροδρόμια. Μερικές φορές τα αεροδρόμια δημιουργήθηκαν και ιδρύθηκαν θα έλεγα κοντά στους πολίτες. Ε, έχουμε 3 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι ζουν πάρα πολύ κοντά στα αεροδρόμια και υποφέρουν από μια ηχητική μόλυνση που ξεπερνά πάρα πολύ συχνά τα 50 δεσιμπέλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά ταχύτατα. Ευχαριστώ. Συνεχίζω τώρα με την κυρία Κριστίν Τεβεράκ. Αλλά δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω στο έδρανό της. Ξέρετε αν είναι εδώ. Αναφέρομαι στην κυρία Ντεβεράκ. Δεν είναι εδώ. Έχουμε τώρα πάρα πολλούς συναδέλφους που θα ήθελαν το λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Θα δώσουμε το λόγο σε εννέα συναδέλφους, δυστυχώς όχι σε περισσότερους γιατί έχουμε μείνει πίσω. Κυρία Λάγκε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω την, ε, ότι η αρμοδιότητα της Κομισιόν για τον έλεγχο και την αναστολή ε, των μέτρων όπως απαγόρευση πτήσεων ακυρώνεται. Αυτό δεν θα ήταν σύμφωνο με την επικουρικότητα. Τέτοιες, ε, τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να ελαμβάνονται μόνο από τις εθνικές αρχές. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όμως ε, που αφορούν την εξισορρόπηση των συμφερόντων και αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Ε, βλέπω ότι ε, μέτρα μετριασμού μπορεί να λαμβάνονται αν δεν επηρεάζεται η χωρητικότητα του αεροδρομίου. Αυτό νομίζω ότι δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του θορύβου και δεν το δεχόμαστε. Ο συνάδελφος Τσέμκε. Χωρίς μικρόφωνο όμως. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τρίτη έκθεση, δηλαδή την έκθεση που σχετίζεται με τις υπηρεσίες εδάφους. Νομίζω ότι ήταν η πλέον αφιλεγόμενη έκθεση κατά τη διάρκεια της συζήτηση. Φαίνεται ότι θα ήταν υποφελές το άνοιγμα της αγοράς για τους επιβάτες. Όμως ανακύπτει το εξής θεμελιώδη ζήτημα. Αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να, να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια για τις επτήσεις και για τους επιβάτες. Ε, ο Αυξημένο ανταγωνισμό δεν πρέπει να συνεπάγεται μειωμένη ασφάλεια και άρα διατυπώνω το εξή ερώτημα προς τον εισηγητή. Έχετε ε, συμπεριλάβει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να, την, ε, θέματα ασφαλείας. Ε, ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Τώρα ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Δύο θέματα θέλω να θέσω. Καταρχώς να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα των χρονοθυρίδων για τα περιφερειακά αεροδρόμια που συνδέονται με τα μεγάλα κεντρικά αεροδρόμια, κομβικά αεροδρόμια. Εγώ προέρχομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Πάρα πολύ σημαντικές οι πτήσεις αυτές για τη λειτουργία της οικονομίας μας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Από ό,τι βλέπω εδώ, η οδηγία του 2002 η οποία προέβλεπε για μία νέα κατηγορία δεν εφαρμόζεται σε ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, κάτω των 15.000 κινήσεων από προσγειώσεων και το αεροδρόμιο ε, George Best είναι, κάτι το, είναι ένα αεροδρόμιο που υπόκειται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και αυτό δημιουργεί επιμέρους προβλήματα. Θα ήθελα να δω λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μπορεί να κάνει. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ. Οι υπηρεσίε εδάφου ε, στα αεροδρόμια δείχνουν ε, καθαρά ποιε είναι οι επιπτώσει τη απελευθέρωση. Απολύσει, ε, έχουμε χαμηλότερου μισθού για του νέου εργαζομένου, περικοπή των μισθών ή μια αύξησή του σε σχέση με τον πληθωρισμό, περισσότερε συμβάσει μερική απασχόληση, επιδείνωση των δεξιοτήτων καθώ και των συστημάτων κατάρτιση και άρα υποβάθμιση των υπηρεσιών εδάφου. Ιδού τα θαύματα τη απελευθέρωση. Τα γνωρίζει αυτά η Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις μελέτες ε, που έχει κάνει η ίδια και για να το διορθώσει, ε, για να προχωρήσουμε, τι κάνει. Όχι, δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ε, επιδεινώνει και εμβαθύνει την απελευθέρωση για να αυξήσει την κερδοφορία. Δεν υπάρχουν όρια στον καπιταλισμό. τα έκαναν τα πάντα για να εντατικοποιήσουν ακόμη περισσότερο την εκμετάλλευση. Και αυτό ισχύει για τους επιβάτες, διότι από αυτά τις αποφάσεις εξαρτάται η ασφάλειά τους. Ε, πρέπει να συνεχίσουν. Κόβεται το μικρόφωνο το ομιλητή. Έχει το λόγο ο κύριος Μπρόνς. Νομίζω ότι είμαι σε επίπεδο αρχής κατά της κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά προτιμώ όταν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία να είναι με τη μορφή κανονισμού και όχι με τη μορφή οδηγίας. Η οδηγία η παλαιότερη του 2002 ήταν αρκετά κακή θα έλεγα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων. Η προτινόμενη νομοθεσία θα προσφέρει περαιτέρω φιλοθεροποίηση. Αυτό σε επίπεδο λογιστικό καλό είναι. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε να κάνουμε με εργασίες στον τομέα της ε, επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, στον έλεγχο ασφαλείας, ε, στις υπηρεσίες εδάφους, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορούμε να το διασφαλίσουμε χωρίς να διασφαλίσουμε ε, την συνέχεια της παροχής υπηρεσίας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μείωση των αμοιβών των εργαζομένων και μείωση του επίπεδου των υπηρεσιών. Ο κύριος Νικουλέσκου έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που ενδιαφερόμεθα πολύ για τους αερολιμένες και τις υπηρεσίες εδάφους η συζήτηση ήταν ενδιαφέρουσα, ήταν καλό που είναι και ο Επίτροπος παρόν. Για να δούμε τώρα τις κρατικές ενισχύσεις για τους αερολιμένες όμως. Πρόκειται για τις ε, ποιοτικέ παροχές υπηρεσιών στα αεροδρόμια και τι προσφέρουν στους επιβάτες οι πάροχοι. Δεν είναι επαρκής η προσφορά, κάποια αεροδρόμια πρέπει να κλείσουν και αυτό έχει επιπτώσεις και στους διάφορους ε, τόπους και περιοχές όπου βρίσκονται οι αερολιμένες. Ε, υπήρξε πρόβλημα και με τη Ρουμανία και το αεροδρόμιο. Πρέπει να σκεφτόμαστε και το μέλλον των αεροδρομίων όταν συζητούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάλτεμπαχ έχει το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 20 ε, χρόνια εσωτερικής αγοράς γιορτάσαμε με πολλά θετικά για τους λαούς της Ευρώπης. Στη, στα θέματα τα εργασιακά πρέπει να βελτιωθούν αρκετά και αν βάζουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, δυστυχώς από την οδηγία σας, την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες εδάφους δεν βλέπω τέτοια βούληση. Ε, η αναγκαστική απελευθέρωση δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα για τους εργαζομένους και αυτό το είπαν αρκετοί συνάδελφοι σήμερα δεν φοβούμεθα μόνο, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μισθολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Και όχι μόνο οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θίγονται. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα που θα υποστεί ε, ζημία. Οι καταναλωτές με τη χειρότερη απασχόλη, ε, εκπαίδευση των ε, εργαζομένων. υπονομεύεται η ασφάλεια των επιβατών. Επίσης θετικό για τις επιχειρήσεις δεν βλέπω επίσης διακοπή. Εξαντλήσατε το χρόνο σας. Η κυρία Κλάις έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πολλά μετράμε σήμερα το θόρυβο σε δεσιμπέλ, αλλά οι επιπτώσεις ε, ε, απευθείας άμεσα στον άνθρωπο δεν μετρούνται εύκολα. Ε, όσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος, τόσο πιο πολύ ευαισθητοποιούμεθα και τόσο πιο πολύ αυξάνεται το στρες. Η είναι σημαντικό οι θυγόμενοι να συμμετέχουν στη λήψη των μέτρων, να εισακούονται. Ε, θα πρέπει αυτό να μείνει στα, χέρια των τοπικών αρχών ε, που ξέρει τις ιδιαιτερότητες κάθε αερολιμένα. Οι επιπτώσεις του θορύβου είναι σε τοπικό επίπεδο, άρα και οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται επιτόπου μαζί με τους ενδιαφερομένους και θυγωμένους ε, θα πρέπει να βρεθούν εξατομικευμένες λύσεις για τα προβλήματα του θορύβου και να να ισχύσουν τελεσίδικα. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία διαμεσολάβησης. Ε, δεν μπορεί αυτή να έρεται από την Κομισιόν. Δεν μπορεί να ε, Διακοπή. Η κυρία Τσίτα Γκουρμάη και κλείνει έτσι ο γύρος της διαδικασίας Catch the Eye. Το μικρόφωνο σας κυρία Γκουρμάη. Okay, fine. Είναι σαφές ότι η πρόκληση που θέτουν τα αεροδρόμια σε μια αγορά ανταγωνιστική πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σχετικά με τις υπηρεσίες εδάφους θα συμφωνήσω με, την με τις απόψεις της πολιτικής μου ομάδας και της αρμόδιας επιτροπής για την απόρριψη της πρότασης δεν προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι προηγούμενες εμπειρίες μας έχουν δείξει ότι τέτοιου είδου ελευθεροποιήσει οδηγούν πάρα πολύ απλά στη λεγόμενο μισθολογικό dumping και ε, στη μείωση των επιπέδων κοινωνικής προστασίας. Ε, έχουμε επιμακρόν ζητήσει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει. Κυρία Γκορμάη, εξαντλήσατε το χρόνο σας. Κλείσαμε τον μεγάλο αυτό κατάλογο ομιλητών. Ε, δυστυχώς ε, μου είναι δυσάρεστο εγώ να μην ανταποκρίνομαι σε όλα τα αιτήματα της μπλε κάρτας επίσης και να μην δίνω το λόγο σε περισσότερους συναδέλφους και στα πλαίσια του Catch the Eye αλλά αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κάλλας, ο οποίος θα απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ακούσαμε τόσες πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και παρεμβάσεις και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη ζωηρή συζήτηση. Δύσκολα μπορώ να σχολιάσω ε, όλες επιμέρους ε, λεπτομέρειες ε, και ούτως ή άλλως είχαμε ευκαιρίες να σαντηθούμε στην Επιτροπή Μεταφορών με πολλούς βουλευτές ε, και μετήχαμε όλες, όλες αυτές τις συζητήσεις και εξάλλου μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε αυτά τα ζητήματα. Εάν αυτό ε, αποφασίσετε φυσικά να συνεχιστεί η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω ότι προφανώς ε, είναι μετριοπαθής η πρόταση. Το πακέτο είναι μετριοπαθές ε, γιατί δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Σίγουρα δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των αερολιμένων και να λύσουμε όλα τα προβλήματα στο εγγύς μέλλον. Βλέπετε ότι στην Ευρώπη ούτως ή άλλως οι πτήσεις συμπιέζονται κυρίως στο κέντρο της Ευρώπης και άρα είναι επιτακτική η ανάγκη να δράσουμε για αυτά τα αεροδρόμια. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ως προς ε, τα θέματα κοινωνικής προστασίας, εγώ ξεκίνησα με τις διαπραγματεύσεις ε, σε μία συνεδρίαση με εκπροσώπους ε, των συνδικαλιστικών οργάνων κατά κάποιο τρόπο ε, νομίζω αποκομίσαμε εντυπώσει σε σχέση με το τι θα συνιστούσε μια ε, ε, ισορροπημένη πρόταση και υπάρχουν περισσότερες διατάξεις σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία σε αυτή τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πραγματικά είναι ισοσκελισμένη η πρόταση αλλά και με διότι μας, με ρωτούν όλοι οι συνάδελφοι τι σημαίνει πλήρης απελευθέρωση. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης μπορούμε να προσθέσουμε διαδρόμους προσγείωσης απογείωσης, νέες χρονοθυρίδες και ούτω καθεξής. Ε, ξέρετε, ε, υπάρχουν πολλές καλές ιδέες ε, από όλες τις πλευρές. Είμαι πεπισμένος πάντως ε, πως είναι μάλλον μετριοπαθές το περιεχόμενο της ε, πρότασης. Ε, τώρα τον επιμείνουμε να περάσει η πρόταση πάση θυσία. δεν μπορώ να κάνω εγώ λόμπινγκ και να ασκώ πίεση για να γίνει αυτό. Αυτή είναι δική σας δουλειά. Πρόκειται για πολιτική απόφαση και δεν πρέπει πρέπει να αντιληφθείτε ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων. Δεν μπορείτε αλλά να επιλέξετε κάποια μέτρα και γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολιτική απόφαση. Αν δεν περάσει το πακέτο δεν θα περάσει. Ακούσαμε διάφορα στοιχεία κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το οποίο θα ήθελα να κάνω πιο συγκεκριμένα ε, και διεξοδικά σχόλια αλλά υπάρχει και ο χρονικός περιορισμός και δεν θέλω να υπερβαίνω το χρόνο αλλά αυτά που ακούσαμε για τις νυχτερινές επτήσεις αυτό είναι τελείως πώς να το πω δεν καταλαβαίνω πώς το ε, ε, σκεφτήκατε καν κύριος Κόλιτσεκ μας έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ότι μπορούμε να οργανώσουμε τις χρονοθυρίδες και τη διαχείριση των αεροδρομίων με εντελώς διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιώντας το ΣΥΖΑΡ και τις νέες τεχνολογίες. Ναι, ναι, είναι εφικτό όμως τα κράτη-μέλη επέλεξαν διαφορετικό τρόπο για να βελτιώσουν τη λειτουργία των υποδομών, κυρίω για τι υπηρεσίε εδάφου και εμεί ακολουθούμε την πρόταση των κρατών μελών. Ωραία. Α δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση του Κοινοβουλίου αύριο και αν δεν τύχει η πολιτική υποστήριξη στο πακέτο θα το αποσύρουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, θα δώσουμε το λόγο τώρα στους ε, τρεις ε, εισηγητές. Νομίζω ότι οι παρόντες συνάδελφοι λόγω ακριβώς του πλούτου της ε, συνεδρίασης που προηγήθηκε, τη συζήτηση που προηγήθηκε. Θα τους δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να κλείσουν τη συζήτηση. Θα είμαστε έμβαση περιπτώσει λιγότερο αυστηροί γιατί ήταν πάρα πολλές οι, οι παρεμβάσεις των βουλευτών και πρέπει να δώσουν απαντήσει. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Τσασάντα, έναν από τους συζητητές αυτής της πολύ σημαντικής συζήτησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος στα σχόλιά μου για να απαντήσω στις πιο συχνές ερωτήσεις. Γενικά, η συζήτηση αυτή έδειξε πόσο μας δυσκόλεψε το θέμα, γιατί ξαφνικά φαίνεται από τη συζήτηση ότι η μεγαλύτερη φιλελεύθερη στην αίθουσα είναι η συντηρητική και ένας φιλελεύθερος που εκπροσώπησε την ομάδα των φιλελευθέρων αποδεικνύεται πολύ συντηρητικός, υπερβολικά συγκρατημένος. Γι' αυτό ε, χάρηκα που επεξεργαστήκαμε πολλές ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και όταν πάει στην Επιτροπή Μεταφορών πάλι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας για τις συμβιβαστικέ. Πολλά επιχειρήματα αναφέρθηκαν. Ο συνάδελφος Λιμπεράτσκι που έφυγε μίλησε για την παραγωγικότητα ως επιχείρημα. Βασικό επιχείρημα κατά του εγγράφου. Τι είναι όμως η παραγωγικότητα πραγματικά. Όταν κάποιος ε, δεν έχει πέντε λεπτά διάλειμμα για να πιει ένα ε, ποτήρι νερό μέσα στο οκτάωρο ή δεν έχει χρόνο να κάνει τίποτε άλλο. Πήγα στο αεροδρόμιο της Ναρίτα πριν από λίγα χρόνια στο Τόκιο και τους ρώτησα ε, ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι ένα αεροδρόμιο πλήρως απελευθερωμένο, χωρίς κανένα εμπόδιο για τους διαχειριστές, για τις εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και να υπογράψουν ε, συμβάσεις ε, μεταξύ αεροπορικών εταιριών και εταιριών υπηρεσιών εδάφους που είναι νέα. Και μετά τους ρώτησε για την παραγωγικότητα. Τι κάνουν οι εργαζόμενοι Οι Ιάπωνες είναι γνωστοί για το σεβασμό που δείχνουν στην εργασία και εξεπλάγησαν που τους ρώτησε τι κάνουν. Έχουν λίγο, αν έχουν ελεύθερο χρόνο, έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο, μπορούν να ξεκουραστούν μπορούν, ή μπορεί να φάνε ή μπορεί να κάνουν κατάλληλη εκπαίδευση δεν ε, έχουν τρεις μέρες υποχρεωτική κατάρτιση. Καταρτίζονται κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα. Ανάλογα με το αν έχουν ελεύθερο χρόνο ή όχι. Το θέμα της προστασίας και της ασφάλειας ε, που τέθηκε είναι ένα από τα κέρια θέματα στο έγγραφο. Κάθε εταιρεία υπηρεσίας εδάφους που θα πάρει έγκριση σύμφωνα με το κείμενο του κανονισμού θα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι μια εταιρεία ασφαλής που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που αφορούν τα πρότυπα προστασίας. Αυτά είναι τα κύρια θέματα σε σχέση με αυτόν τον κανονισμό. Και τώρα ένα θέμα που αφορά τους ε, συναδέλφους πρασίνους και σοσιαλιστές όπως και τους συναδέλφους από την αριστερά και τους συναδέλφους από το ΕΛΚ επίσης που ενδιαφέρθηκαν για το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και που πολλές φορές αναφέρθηκαν σε σημαντικά κοινωνικά θέματα, εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ε, αυξάνοντας το αίσθημα ασφαλείας. Διακόπη, έκλεισε το μικρόφωνο. Σαν εισηγητής επίσης έχει το λόγο τώρα ο κύριος Αλλά συνεχίζει, ο κύριος Ζασάντα ο κ. Σουτζίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρουσιάσει μια κάποια σύνθεση μέσα σε ένα τόσο λίγο χρόνο και αυτό απεδείχθη από την παρέμβαση Ζασάντα. Πάντω θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου, οι οποίοι προσπάθησαν να συνεισφέρουν στη συζήτηση αυτή να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και του συμβούλους μας και υπαλλήλους που πήραν μέρος στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για τα θέματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί. Το πρώτο, για τον κίνδυνο να επηρεάσουμε με, ε, το, τη ρύθμιση που προβλέπεται για τις χρονοθυρίδες την ε, την σύνδεση ορισμένων περιφερειοκών με τα κομβικά αεροδρόμια. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να ελέγξουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο πολλούνται τα σλότς έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η συνδεσιμότητα των διαφόρων περιοχών με τα κεντρικά κομβικά αεροδρόμια. Εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασώσουμε αν θέλετε ε, τις περιφερειακές και νησιωτικές μάλιστα περιοχές. γενικά το θέμα των σειρών σαν παράδειγμα το οποίο έτσι όπως προβλέπετε θα πρέπει να αντικαταστήσει κάποιες αρχές ε, οι οποίες ισχύουν μέχρι τώρα ε, θα πρέπει όλα αυτά να ρυθμιστούν νομικά πλέον για να διασφαλιστεί η επιθυμητή συχνότητα σύνδεσης. Είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην σημερινή ε, συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά λόμπι τα οποία ενδιαφέρονται. Έχει υπάρξει έκφραση ενδιαφέροντος από συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και από συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και αυτό δεν θα πρέπει να μας αποτρέψει από το να εξυπηρετήσουμε πριν από οτιδήποτε άλλο το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα να καλέσω όλους λοιπόν σχετικά με τις χρονοθυρίδες να στηρίξουν τον νομικό ορισμό των χρονοθυρίδων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια νομική πλαισίωση του καθεστώτος των χρονοθυρίδων και της χρήσης των χρονοθυρίδων να αναγνωριστεί ο, ο χαρακτήρας δημοσίου συμφέροντος τον οποίο έχουν οι χρονοτηρίδες. Και θα ήθελα εδώ τώρα να πω αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του κυρίου Κάλλας, ο οποίος έθεσε συγκεκριμένα θέματα με πολύ θαραλέο τρόπο, με κάθε ειλικρίνεια θα πρέπει να του πω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας σεβασμός της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία εκφράστηκε υπέρ δύο από τις προτάσεις τις οποίες έκανε η Επιτροπή σήμερα. Δεν μπορεί να αγνοηθεί η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρξει σεβασμός στην άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον οποίο οφείλεται στην ψήφο εμπιστοσύνη στην οποία λάβατε στην αρχή της εντολής σας και στην αρχή της εντολής της Επιτροπής του κ. Μπαρόσο. Δεν έχετε άλλο χρόνο λέει ο κύριος Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κύριο Λάιχτφρεντ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την έκθεση για το θόρυβο δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Χαίρομαι γιατί κατέστη σαφές προς όλους και όλοι δέχονται ότι η προστασία της υγείας των ε, ανθρώπων ε, υπερέχει των οικονομικών συμφερόντων. Όλοι συμφωνούμε και έτσι θα συμπεριφερθούμε και στην ψηφοφορία. Ε, τώρα, για, επειδή έχω λίγο χρόνο, δύο λόγια για τις υπηρεσίες εδάφους. Κύριε Επίτροπε, η πολιτική σας και η, συν, η πραγματικά ε, έχουν, ε, προσκρούν στα ε, συμφέροντα των ανθρώπων που έχουν πια βαρεθεί το νέο φιλελευθερισμό και το ρόλο που έπαιξε στην χρηματοπιστωτική κρίση που σημαίνει μειωμένη ασφάλεια, μειωμένα εισοδήματα, μειωμένες θέσεις εργασίας, απασχόληση και στο μέλλον αν ακολουθήσουμε έτσι τότε θα ε, έχουμε ε, ε, πρόβλημα διότι τα, η ενιαία αντιμετώπιση των αεροδρομίων ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες από οτιδήποτε δεν οδηγεί πουθενά. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν δει ανθρώπους που διαδηλώνουν ερχόμενοι από πολλές, πολύ μακρινές περιοχές για να διαμαρτυρηθούν και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τους αγνοούμε. Ε, υπάρχουν άνθρωποι δραστήριοι, ε, άνθρωποι που μας ψηφίζουν και που θα ε, καταπολεμήσουν στην πράξη τέτοιου είδους κανονισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντάλεν, διαδικαστικό. Ναι κύριε Πρόεδρε. Διαδικαστικό για προσωπικού λόγους. Αναφερθήκατε και στους ε, συνεργάτες ε, της Επιτροπής. Κοιτάξτε, εγώ εξέφρασα μια πολιτική άποψη γύρω από το θέμα αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν στα πλαίσια αυτής της συζήτηση να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση και φυσικά να λάβουμε υπόψη μας και τα θέματα της απασχόλησης. Ελάτε τι γίνεται στο Skip Call. Αυτό δεν ήταν διαδικαστικό κύριε Βαντάλε. Αυτό είναι μια άποψη την οποία δικαιούστε να έχετε, αλλά δεν ήταν για να την πείτε εδώ. Λοιπόν, ήταν μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. και ιδιαίτερα για τους αυτό φάνηκε και από τους συναδέλφους ε, που έμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης τιμά την ε, Ολομέλεια και το Κοινοβούλιο η παρουσία όλων αυτών των συναδέλφων Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για την παρουσία του και τις απαντήσεις του. Η ψηφοφορία θα γίνει, έκλεισε η συζήτηση, αύριο το μεσημέρι, τη 12η μεσημβρινή. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης να δώσουμε λίγο χρόνο για να υπάρξει η θα έλεγα αλλαγή της θέσης των επιτρόπων ή έχουμε να κάνουμε με τη σύσταση της κυρίας Ποδήματα για την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ένα άλλο θέμα υψηλής σημασίας και ενδιαφέροντος και για το συγκεκριμένο θέμα έχουν εγγραφεί ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι, πολύ περισσότεροι από ό,τι συνήθως. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Ποδήματα. Έχετε στη διάθεσή σας κυρία Ποδήματα έξι λεπτά. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπως εσείς πιστεύετε. Θέλετε τέσσερα λεπτά για να παρουσιάσετε